Αρχίζουμε με την ψηφοφορία. Par, euh, euh, Αρχίζουμε πρώτα απ' όλα με την έκθεση της κυρίας Στίφλερ. Έχουμε δύο τροπολογίες. Τροπολογία αριθμός 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ηλεκτρονική ψηφοφορία επί του συνόλου της έκθεσης. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Έληξε η ψηφοφορία. 26 ψήφοι υπέρ. Ναι, ναι, γράφει 24 στην οθόνη, αλλά δύο δεν έχουμε την ε, κάρτα μας. Λοιπόν, ψηφίζουμε τώρα την ε, έκθεση νομοδότης της Κατρίν Γκρέζ. Αρχίζουμε πρώτα απ' όλα με την ε, τροπολογία 2 του κυρίου Ντέβα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Λίγη ψηφοφορία. Απορρίπτεται με 12 προς 15. Συμβιβαστική τροπολογία α. Υπέρ. Καλά. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 3. Όχι, καταπίπτει. Καταπίπτει η 3. Τροπολογία 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Η ηλεκτρονική επελήθευση. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Λίγη ψηφοφορία. 11 προς 16 απορρίπτεται. Τροπολογία 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 7. Υπέρ. Θέλετε ηλεκτρονική επαλήθευση της 6. Πολύ καλά. Αρχίζει η ψηφοφορία για την ηλεκτρονική επαλήθευση της τροπολογίας 6. Ψηφίσατε όλοι. Λίγη η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Τροπολογία 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση αρχίζει η ψηφοφορία Λίγη ψηφοφορία και εγκρίνεται η τροπολογία. Τροπολογία 10. Υπέρ. Κατά. Εποχές. Απορρίπτεται. 11. Όχι. 12. Υπέρ. κατά, αποχές εγκρίνεται. 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 14. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 15. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 16. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική ψηφοφορία Β. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Είκοσι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία σε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 24 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση. Αρχίζει η ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 25 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 25 υπέρ, 20, 26 26 λοιπόν. 26 υπέρ, κατά, εποχές, απορρίπτεται. Ηλεκτρονική επαλήθευση της 26. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Λίγη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 27. Καταπίπτει. 28. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 29. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 10, χωριστή ψηφοφορία. Πρώτο μέρος, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. ηλεκτρονική επαλήθευση του δεύτερου μέρους της συμβαστικής ΔΕΛΤΑ. Αρχίζει ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Λίγη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 14 προς 12. 34. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 35 υπέρ, κατά, αποχές, η ηλεκτρονική επαλήθευση. Αρχίζει ψηφοφορία για την 35. Ψηφίσατε όλοι. Λίγη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Προφορική τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 36 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 37 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 38 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τη γνωμοδότηση έτσι όπως την ε, τροποποιήσαμε. Αρχίζει ψηφοφορία, ψηφίσατε όλοι. Λίγη ψηφοφορία. εγκρίνεται με 15 προς 11. Θα περάσουμε τώρα στην ψηφοφορία της επόμενης έκθεσης. Συντάξτε γραμματότητα η κυρία Μισελ Στίφλερ. Πρώτη τροπολογία. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δύο. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε μαζί τις τρεις τροπολογίες, 3, 4, 5, υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται, προφορική τροπολογία 1, υπέρ κατά αποχές Ηλεκτρονική επαλήθευση. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Λίγη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Τροπολογία 7. Υπέρ.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 εποχές απορρίπτεται 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται λεκτή ηλεκτρονική ψηφοφορία για την γνωμοδότηση έτσι όπως τροπολογήθηκε υπέρ. Ε, συγγνώμη, αρχίζει η ψηφοφορία. «26 προς 1. Μία εγκρίνεται». περάσουμε στο σημείο 14 της ημερήσιας διάταξης για το δημοκρατικό έλεγχο του προγραμματισμού στο πλαίσιο της νομοθεσίας που διέπει την αναπτυξιακή πολιτική. Έχουμε ήδη λάβει από την Επιτροπή το πρόγραμμα μετανάστευση και άσυλο έγγραφο στρατηγικής 211-213 για την χρηματοδότηση της ε, ανάπτυξης και συνεργασίας. Εξετάστηκε το εν λόγω έγγραφο από την ομάδα εργασίας ΣΕ και ζητώ στην εισηγήτρια να παρουσιάσει τις συστάσεις και τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξε η ομάδα εργασίας της. Η κυρία Κέλλερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Θα σας παρουσιάσω τα συμπεράσματα της ομάδας εργασίας C όσον αφορά τα θεματικά, το θεματικό πρόγραμμα για τη μετανάστευση και το άσυλο. Ήταν καρποφόρα ανταλλαγή απόψε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανταλλάξαμε και επιστολές, κάποιες ερωτήσεις, απαντήσεις και τα συμπεράσματα τα βλέπετε στο έγγραφο αυτό που διενεμήθη στις θέσεις σας. Να σας παρουσιάσω λοιπόν τα βασικά συμπεράσματα τα οποία συναγάγαμε. Πρώτα απ' όλα έχουμε κάποιες επικρίσεις. Δηλαδή θεωρούμε αρνητικό το ότι δεν βλέπουμε τους στόχους που εμπεριέχονται ούτε τα κριτήρια να αντικατοπτρίζονται πλήρως στον προϋπολογισμό. Όπως ξέρετε το άθρο 20 του σχετικού κανονισμού αναφέρει ότι τα έγγραφα θεματικής στρατηγικής θα πρέπει να αναφέρονται σε ενδεικτικά οικονομικά ποσά και εν γέννη και κατατομής προτεραιότητας Οπότε πρέπει να προβλέπετε ένα κονδύλιο προπολογισμό για το θεματικό πρόγραμμα. Αυτό είναι το κανονικό. Και οι πέντε τομεί προτεραιοτήτων εδώ είναι η ισχυροποίηση της, ε, των συνδέσεων μεταναστεύσεως και ανάπτυξη. Θα πρέπει να οργανωθεί καλύτερα νόμιμη μετανάστευση, να καταπολεμηθεί η παράνομη μετανάστευση, Τέταρτον, προστασία των μεταναστών. Τέταρτον, να προωθηθεί το άσυλο και διεθνή προστασία. Εδώ θα θέλαμε να βλέπουμε πόσα χρήματα θα διατεθούν και ποια χρήματα πάνε σε ποιο τομέα προτεραιότητα. Δυστυχώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ήταν σε θέση να μα δώσει τι ενδείξει. Έλεγε ότι χρειάζεται ευελιξία να μπορεί να μετακινεί τα διάφορα ποσά. Εμείς είπαμε ότι για να υπάρχει ευελιξία θα ήταν σημαντικό να υπάρχει ένας κανονικός προϋπολογισμός, ο οποίος προϋπολογισμός θα μπορεί να αντιμετωπίζει αλλαγές, χρειάζεται όμως ένας σχεδιασμός στα πλαίσια ενός προϋπολογισμού. Μας διαβεβαίωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι το, για κάθε μία προτεραιότητα θα δίδεται ανάμεσα στο 10 με 30% του ποσού. Έχουμε κάποιον αριθμό, έχουμε κάποιο αριθμητικό στοιχείο, έστω και αυτό. Συστήνουμε να ακολουθήσουμε να συμφωνήσουμε επαγρυπνώντας την περαιτέρω εφαρμογή του προγράμματος, ούτως ώστε να εξασφαλίσουμε ότι κάθε τομέας προτεραιότητας θα πάρει το μερίδιο που του αρμόζει και δεν θα παραμελείται. Αυτά λοιπόν για τα κονδύλια, για τη χρηματοδότηση. Δεύτερον, υπήρχαν κάποιες αφιβολίες όσον αφορά την συμβατότητα. Τα θεματικά προγράμματα, 90% των δαπανών διατίθεται βάσει των κριτηρίων όντα. 10% δεν μπαίνει σε αυτό το, δεν εντάσσεται σε αυτό τον τρόπο κατανομής, όντα. Η ενδιάμεση αναθεώρηση που έγινε έδειξε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδότησε 12 από τα 60 προγράμματα, οπότε αυτό καλύπτει το 11,6% από το 2007 μέχρι το 2009 τη συνολική χρηματοδότηση και βάσει των στοιχείων που είχαμε στη διάθεσή μας, θεωρήσαμε ότι ήταν ανέφικτο να διαπιστώσουμε κατά πόσο έχει πληρωθεί το κριτήριο το 10% και υπάρχουν και γενικότερα προβλήματα. Δεν υπάρχει κώδικας για μεταναστευτικές δραστηριότητε στα κριτήρια DOC και ήταν δύσκολο για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταρτήσει κατά πόσο μπορούν να ενταχθούν σε αυτό το πλαίσιο ή όχι των συγκεκριμένων κριτηρίων. Συμπεράναμε λοιπόν ότι η αξιολόγηση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ότι μόνο το 0,2% των δραστηριοτήτων που χρηματοδοτούνται από τα DCI θεματικά προγράμματα δεν μπορούν να ενταχθούν στο πλαίσιο τάκ Καλό ποσοστό, αλλά επικρατεί ένα συνέστημα ανασφάλειας, αμφιβολία. Ανησυχούμε πολύ λοιπόν για την αβεβαιότητα που επικρατεί τι εντάσσεται στο σωστό πλαίσιο και τι όχι, στο πίσω ντό και τι όχι. Και ανησυχούμε για μια από τις βασικές δραστηριότητες στους γεωγραφικούς τομείς προτεραιότητας. Πρόληψη και έλεγχος παράνομης μετανάστευσης. Εκεί μπορεί να πει κανεί αυτό πώς σχετίζεται με την εκρίζωση της στόχιας, πώς σχετίζεται με τα κριτήρια DAC και ο μεθοριακός έλεγχος των διαφόρων χωρών είναι κοινοβουλευτική ε, απασχόληση, αν θέλετε, αρμοδιότητα και δεν είναι ξεκάθαρο σε ποιε δραστηριότητε φορέων γίνεται η ε, χρηματοδότηση. Στην ενδιάμεση αναθεώρηση λέει ότι αν δίνονται χρήματα σε μια οργάνωση, ε, επειδή δεν ασχολείται με ανάπτυξη, ίσως όσον αφορά δεν μπορεί να ενταχθούν στους στόχους της χιλιατίας. Λοιπόν, και ποιε δραστηριότητε μπορούν να χρηματοδοτούνται σωστά και να μπορούν να ενταχθούν στου στόχου τη χιλιετία, γιατί βεβαίω είναι σημαντική α, μέρημνα αυτή τη Επιτροπή. Θα ήθελα λοιπόν να πω ότι υπάρχουν κάποιες ελλείψεις. Δεν υπάρχει συνεχή όσον αφορά την ανάλυση των βασικών διεθνών προκλήσεων και τις απαντήσεις από την άλλη που προτείνονται ε, στο πρόγραμμα πλαίσιο. Βλέποντα αριθμού, βλέπουμε ότι η διεθνή μετανάστευση είναι σε κλίμακα νότου προ νότον. Και αν δείτε μετανάστευση προ την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι μεγαλύτερε ομάδε μη Ευρωπαίων μεταναστών ήταν πολίτες το 2004 από την Ασία, Βόρεια, Κεντρική και Νότια Αμερική. Ενώ εδώ δίνουν προτεραιότητα σε μετανάστευση από Αφρική, κυρίως Βόρεια Αφρική και υποσαχάρη Αφρική προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και περιθωριοποιεί μεταναστευτικές ροές από Λατινική Αμερική καθώς και μεταναστευτικές ροές από αναπτυσσόμενες χώρες προς αναπτυσσόμενες χώρες. Το βλέπουμε ως πρόβλημα αυτό και φαίνεται να εστιάζεται περισσότερο λοιπόν το, το στρατηγικό αυτό πρόγραμμα στα μεταναστευτικά προβλήματα που αντιμετωπίζονται και είναι εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ενδιάμεση αναθεώρηση συνέστησε η μετανάστευση νότου προς νότο να παίξει μεγαλύτερο ρόλο στο θεματικό πρόγραμμα. Επίσης θα θέλαμε να πούμε ότι είναι από τους στόχους η μετανάστευση στο νότο του προγράμματος και αυτός ο τομέας χρειάζεται συγκεκριμένη στρατηγική ώστε να έχουμε προσμετρήσιμα αποτελέσματα. Παραδείγματο χάρη, η ενδιάμεση αναθεώρηση πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συσφίξει τη συνεργασία με φορείς περιφερειακή συνεργασίας, με εντολή για οικονομική περιφερειακή συνεργασία συμμεταμονούμενων και θεμάτων μετανάστευσης νότου-νότου. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το λαμβάνει υπόψη της και το προωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανθρώπινα δικαιώματα, πώ εντάσσονται σε όλε πολιτικέ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκεί λέει ότι η συμπερίληψη ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλε πολιτικέ θα πρέπει να λάβει χώρα, σε όλα τα προγράμματα, σε όλε τι δραστηριότητε. Αλλά μα έλειπε κάποια στρατηγική σχετικά με το πώ ακριβώ θα εφαρμοστεί αυτό, πώ τα ανθρώπινα δικαιώματα θα ενταχθούν στι πολιτικέ και πώ θα δοθεί ιδέουσα προσοχή. Το ίδιο και για την ισότητα των φύλων, πώ εντάσσεται στι διάφορε πολιτικέ. Τι ευαισθητοποίηση υπάρχει Χρειάζεται θέματα ισότητα των φύλων και στον τομέα τη μετανάστευση να λαμβάνονται υπόψη, όπω και άλλου τομεί, αλλά λείπει κάποια στρατηγική πώ όλα αυτά θα λαμβάνονται υπόψη όταν θα εφαρμόζονται τα συγκεκριμένα προγράμματα και δραστηριότητε. Υπήρχαν και άλλα σημεία που συζητήσαμε, αυτά ήταν τα βασικά μα πορίσματα όμω. Και στο τέλο, όπω συζητήσαμε και την περασμένη φορά, προτείναμε να μην απορριφθεί το πρόγραμμα, αλλά να το παρακολουθούμε εκ του σύνεγγυ από Το πώ υλοποιείται πώς εκτελείται. Να δούμε πώς καλύπτονται οι ανησυχίε μας. Κυρίως γιατί κάποιες από τις ανησυχίε που μόλις σας ανέφερα εκφράστηκαν και στην περασμένη ενδιάμεση αναθεώρηση. Άρα τίποτα δεν είναι καινούριο και δεν πρέπει να δημιουργεί έκπληξη και νομίζω ότι θα πρέπει με άγρυπνο όμα να παρακολουθούμε τα τεκτενόμενα. Αυτά είναι τα απορίσματα. Ευχαριστώ που με ακούσατε. Ευχαριστώ πολύ. Δίνουμε το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στον κύριο Μάρτιν Πένιγκτον δίνουμε Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και τους εισηγητές για τις ε, σαφείς εξηγήσει για τα θέματα που μας απασχολούν. Ε, θεώρησα ότι αυτό ήταν πολύ ενδιαφέρον διότι επικεντρώνεται σε βασικά θέματα και διότι ε, από πλευράς ε, παρουσιάσεως για το διάλογο για το που βρισκόμαστε νομίζω ότι η κατάσταση ήταν πολύ σαφής. Ε, υπάρχουν ένα-δύο θέματα που αναφέρονται στην εφαρμογή του προγράμματος και που μπορέσαμε να συμφωνήσουμε. Ε, καταρχάς ορισμένα έρχονται εκ των υστέρων διότι ε, έχουμε χάσει την ευκαιρία να διατυπώσουμε προτάσεις και δεν γνωρίζουμε ποιες είναι οι, ποιοι είναι οι οργανισμοί που θα το προωθήσουν. Οπότε, ε, στην ε, Επιτροπή αυτή πρέπει να το κοιτάξουμε. Ε, πρέπει να σας ενημερώσω ότι καταρχήν ε, συμφωνήσαμε και συζητήσαμε για τους πέντε τομείς κατά προτεραιότητα και ε, είχαμε προτεραιότητες. Το ένα θέμα ήταν ότι προσπαθήσαμε να καλύψουμε, ε, καταρχήν ε, να, καταρτήσουμε πέντε προτεραιότητες. Δεύτερον, να καλύψουμε τις πέντε προτεραιότητες μέσω των ε, προγραμμάτων στόχος και θα αποδείξουμε όσο προχωρά το πρόγραμμα ότι εμείς εφαρμόζουμε τους κανονισμούς. Το άλλο θέμα που ήθελα να θίσω ήταν ε, η δυνατότητα αξιολογήσεως την οποία εμείς χρηματοδοτούμε αλλά και η αφαιρεσιμότητα absolutely με συγχωρείτε δυνατότητα να περιληφθεί στο στόχο της χιλιετηρίδας στο κάθε πρόγραμμα ε, μέσα στα πλαίσια των προγραμμάτων και γι' αυτό θα προσέξουμε πάρα πολύ να μπορούμε να σας ενημερώνουμε ε, ε, για το περιεχόμενο αυτών των θεματικών ενωτήτων και το κατά πόσον συνάδουν με το πρόγραμμα γιατί πρέπει να είμαστε πολύ σαφείς. Ευχαριστώ πάντως ε, τον εισηγητή και ε, την ομάδα του διότι νομίζω ότι είναι πάρα πολύ επικοδομητικό να μπορούμε να κάνουμε αυτές τις ασκήσεις. Ευχαριστώ. Συμφωνείτε με την ε, άποψη της εισηγητρίας τότε θεωρώ ότι ε, υιοθετήθηκαν η, ε, η διαδικασία ε, για το, ε, την ενημέρωση σχετικά με την διάσκεψη κορυφής και λίγη το, το θέμα αυτό. Τώρα προχωράμε στο επόμενο θέμα που είναι ε, η έκθεση του κυρίου Κασμάρεξ σχετικά με την αύξηση του αντικτύπου της αναπτυξιακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Και εδώ πρόκειται για ένα πολύ βασικό μέσα για να μπορέσουμε να αυξήσουμε τις δυνατότητές μας διότι στο μέλλον θα πρέπει να αναφερόμαστε σε μηχανισμούς οι οποίοι καταρχήν επιτρέπουν να υλοποιούμε τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ενώσεως αλλά σε συνδυασμό με δάνεια από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και άλλους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς για να καλύψουμε τα επενδυτικά προγράμματα. Θέλω να ε, καλωσορίσω τον κύριο Βόλφκαν Ρόι, στον τον ε, ε, εμπειρογνώμονα της Γενικής Τραπέζης FKV και την εκπρόσωπο του, της ε, οργανώσεως γυναικών καθώς επίσης και στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δίνω λοιπόν καταρχήν τον λόγο εις ε, τον, εις ε, τον εισηγητή κύριο Κασμάρεκ. Η, το φαινόμενο της ε, εφαρμογής ε, των, ε, και υλοποίησης των δανείων είναι πολύ σημαντικό και στηρίζουμε αυτό τον τρόπο χρησιμοποίησης της αναπτυξιακής βοήθειας η οποία αποβλέπει στο να επιτρέψει κάποια μόχλευση ιδίως για τη χώρα μέσων εισοδημάτων και στις χώρες αυτές πρέπει ε, να έχουμε υπόψη μας ότι υπάρχουν πάρα πολλά άτομα που ζουν σε τεράστια ένδια. Πρέπει λοιπόν να ε, συνδυάσουμε τη χρηματοδότηση μαζί με αυτήν της ε, επενδυτικής τράπεζας για να προσφέρουμε πλέον των χρημάτων και μια υποδομή και τεχνική βοήθεια και να κατανείμουμε τους κινδύνους που ε, αντιμετωπίζουν οι επενδύσεις σε αυτές τις χώρες. Από την δικιά μας άποψη, αυτό που είναι σημαντικό εδώ είναι να έχουμε υπόψη μας ότι μιλάμε για νέα χρηματοδότηση, διότι λέμε ε, πάντοτε ότι όλη αυτή η επιπρόσθετοι πόροι πρέπει να είναι μία προσθήκη. Έχουμε λοιπόν την ε, επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια και αυτή πρέπει να ε, χρησιμοποιηθεί χρησιμοποιείται. Πέραν αυτού όμως υπάρχει ε, και επιπρόσθετη χρηματοδότηση είτε μέσω μοχλεύσεως είτε άλλων μεθόδων. Πρέπει όμως αυτό να προσφέρει επιπλέον χρηματοδότηση ε, πέραν της ε, συνήθους. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ο πάντοτε έχει στηρίξει την προσπάθεια αυτή βάσει εις, ε, την έκθεση την οποία είχαμε καταρτήσει σχετικά με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Υπάρχει δηλαδή στήριξη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρέπει όμως να ληφθούν υπόψη και άλλα στοιχεία εξού και γίνεται η συζήτηση σήμερα. Πώς θα προχωρήσουμε. Γιατί ο μηχανισμός αυτός δεν είναι και τόσο καινούριο. Έχει χρησιμοποιηθεί ο δανεισμός επί σειρά ετών με ικανοποιητικά αποτελέσματα, αλλά πρέπει να επιλέγουμε σωστά τους ομολόγους μας και τα προγράμματα που θα χρηματοδοτούμε. Ε, ε, θα πρέπει δε να χρησιμοποιούνται και εμπειρογνώμονες. Θα ακούσουμε τώρα τους, τα μέλη της Επιτροπής, τους εμπειρογνώμονες με συγχωρείτε και ε, τον λόγο θα έχουν ο καθένας για 10 λεπτά. Δίνω πρώτα το λόγο στον κύριο Ρόις. Good afternoon, ladies and gentlemen, um, and members of the parliament. Καλησπέρα κυρίε και κύριοι και μέλη του Κοινοβουλίου. Για μένα είναι χαρά, αλλά και τιμή να έχω τη δυνατότητα σήμερα να μιλήσω σε εσά και να αναφερθώ στη δική μα εμπειρία όσον αφορά τον σχεδιασμό από πλευρά ε, χρηματοπιστωτικού ιδρύματο. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο πιο σύντομο και επακριβή μπορώ και νομίζω ότι μετά θα μπορέσουμε να ακούσουμε τι ερωτήσει, μετά που μπορούμε να συζητήσουμε. α κάνουμε σύντομη εισαγωγή, να σας πω ποιοι είμαστε, η KFW είναι μεγάλη ε, τράπεζα εμπορική που έχει τις περισσότερες επιχειρήσεις εντός Γερμανίας. Προωθούμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, έχουμε ιδιαίτερη, δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στην αλλαγή του κλίματος και στα πλαίσια των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και με τους ιδιώτες πελάτες. Και εκεί είμαστε σαν ε, τράπεζα που χρησιμοποιεί το γερμανικό τραπεζικό σύστημα με μεγάλα ποσά, 75-80% νέες ε, υποχρεώσεις αναλάβαμε, δισεκατομμύρια συγγνώμη, αναλάβαμε πέρσι, τα περισσότερα στη Γερμανία. Εκτός από τη θηρίδα μας στη γερμανική, των επιχειρήσεων εργαζόμαστε και διεθνώς και εκεί έχουμε μια θηρίδα όπου χρηματοδοτούμε, χρηματοδοτούμε προς το εξωτερικό, χρηματοδοτούμε προγράμματα και έργα τα οποία είναι επί εμπορικής με θηγατρική. Την KFW Apex Bank μας. Και έχουμε ε, και ένα υποκατάστημα για αναπτυξιακή βοήθεια, η DG, που ε, προωθεί τον ιδιωτικό τομέα στις αναπτυσσόμενες χώρες. Και έχουμε και την Αναπτυξιακή Τράπεζα, που είναι υπεύθυνη για χρηματοπιστωτική συνεργασία, όπου κυρίως εργαζόμεθα εκπροσωπώντας περισσότερο τη γερμανική κυβέρνηση στις αναπτυσσόμενες χώρες. Αυτό που είναι σημαντικό για να σας δώσω μια φωτογραφία με εικόνα, είναι ότι δρούμε σαν αναπτυξιακή τράπεζα, δεν είμαστε επενδυτική τράπεζα. Τι σημαίνει αυτό. Πρώτα απ' όλα για μας σημαίνει ότι ευθυγραμμιζόμαστε στις ανάγκες του πελάτου. Δηλαδή, ο εταίρος μας είναι πάντα αυτός που οδηγεί. Είτε για σύμβαση για παροχή συμβουλών, είτε για κάποιο έργο. Λαμβάνουμε υπόψη το συμβαλόμενο μέρος και αυτό καθορίζει, το συμβαλόμενο μέρο καθορίζει την ταχύτητα. Και η γερμανική χρηματοπιστωτική συνεργασία ε, γίνεται ανοιχτά μέσω διεθνών διαγωνισμών. Προσπαθούμε να προωθούμε βιώσιμα προγράμματα. Τι σημαίνει αυτό. Εξετάζουμε τις ανάγκες του κάθε τομέα. Προσπαθούμε να επιφέρουμε αλλαγές προωθώντας, βελτιώνοντας το περιβάλλον του προγράμματος το οποίο προωθούμε για να είναι βιώσιμο πέραν αυτού. Προωθούμε και τους συνεργαζόμενους θεσμικούς φορείς, αυτούς με τους οποίους συνεργαζόμαστε. Έχουμε συνοδευτικά μέτρα, εκπαιδεύουμε τους εταίρους μας, τους βάζουμε σωστή θέση, ούτως ώστε να μπορούν να εκτελούν τα προγράμματα, να τα υλοποιούν και να τα χειρίζονται στο μέλλον για μας είναι πολύ σημαντικό να έχουμε συγκεκριμένη ομάδα στην οποία στεζόμαθα. Ομάδες στόχους έχουμε. Θέλουμε να απευθυνόμαστε στους ανθρώπους, να λαμβάνουμε υπόψη βέβαια τις ε, πτυχές που, που χρειάζεται, όπως η ισότητα των φύλων λοιπά στην προσέγγιση και περιβαλλοντικός αντίκτυπος είναι στο επίκεντρο των όσων συζητούμε και εξετάζουμε. Πέρα από την αξιολόγηση περιβαλλοντικών συνεπειών, φροντίζουμε και πιο συγκεκριμένα θέματα του κλίματος. Προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε στο μέτρο του δυνατού, τα λαμβάνουμε όλα αυτά υπόψη. Δηλαδή ότι η ενίσχυση για την οποία είμαστε υπεύθυνοι χρησιμοποιείται αποτελεσματικά. Τι σημαίνει αυτό. Παρακολουθούμε τα προγράμματα από την αρχή. Υποστηρίζουμε την προσδηματία τους. Γίνονται μελέτες ε, βιωσιμότητας. Ε, εξετάζουμε όλες τις στις πτυχές. Κατά την εκτέλεση Παρακολουθούμε αισθανά τι γίνεται. Να είμαστε σίγουροι ότι γίνεται σωστή χρήση των πόρων. Ότι τηρείται το χρονοδιάγραμμα. Και ότι γίνεται σεβαστό και το αρχικό πρόγραμμα χρηματοδότησης. Και εξίσου σημαντικό, στο τέλος του κύκλου του προγράμματος και του έργου, τη στιγμή που λειτουργεί το πρόγραμμα, πάντα κάνουμε τελική αξιολόγηση. Προσπαθούμε να μάθουμε τι πήγε καλά, τι πήγε στραβά ούτως ώστε να μπορούμε στο μέλλον να μάθουμε και να προωθούμε την καλύτερη πρακτική. Σας δίνω λοιπόν τρία σύντομα παραδείγματα προγραμμάτων στα οποία έχουμε συμμετάσχει και αφορά το θέμα του σχεδιασμού. Δύο από αυτά εντάσσονται στη Βόρεια Αφρική, στα πλαίσια Βορειοαφρικής και Μέση Ανατολή. Είμαι υπεύθυνο για αυτή την περιοχή και αυτά τα, αυτές οι διευκολύνσεις έχουν χρησιμοποιηθεί, λειτουργούν καλά, έχουμε αγωγό ε, χορήγησης των πόρων και έχουμε και ένα πρόγραμμα για ένα έργο στην Ουγγάντα για παροχή ύδατος. Λοιπόν, τώρα έχουμε πρόγραμμα για, για την Αίγυπτο, για υδροδότηση και αποχέτευση. Υποστηρίζουμε λοιπόν το πρόγραμμα γιατί. Διότι έχουμε σημαντικές απώλειες υδάτων, υπάρχουν σημαντικά προβλήματα όσον αφορά την ποιότητα του νερού και αντιμετωπίζουμε κεντρικό σύστημα σε αυτούς τους τομείς και θέλουμε να τα αποκεντρώσουμε τα μέτρα και τα αργά. Μιλάμε για υποδομές, βελτίωση ε, της κατάστασης των υδάτων, των υγρών αποβλήτων και αποκέντρωση. Με το πρόγραμμα αυτό ερχόμαστε σε επαφή με τέσσερις κυβερνήσεις στην Άνω Αίγυπτο και γέννη καλύπτουμε πάνω από 50 εκατομμύρια ανθρώπους. Τους περισσότερους στην Ήπεθρο, όπως θα βλέπετε. Και βέβαια, γενικότερο στόχος του προγράμματος είναι η βελτίωση της υγείας του πληθυσμού, να συμβάλλουμε στην προστασία του περιβάλλοντος και των υδατίνων πόρων και τέλος, εξίσου σημαντικό, να προωθήσουμε μεταρρύθμιση του τομέα, να αποκεντρωθεί η παροχή αυτών των υπηρεσιών και το πρόγραμμά μας μάλλον να μπορούν να σταθούν στα πόδια τους οι διάφοροι φορείς που εκτελούν και υλοποιούν το πρόγραμμα επιτόπου. Είναι ένα μεγάλο πακέτο οικονομικό όπου έχει αναφηθεί η ABD και η FD και η KFW. Συμβάλλει σημαντικά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 13 εκατομμύρια ευρώ τεχνικής βοήθειας και αυτό αφορά υποστήριξη μεταρρυθμίσεως του τομέα και την υποστήριξη των εκτελεστικών φορέων για να μπορούν να λειτουργήσουν στο μέλλον αποκεντρωμένα. Πέραν αυτού, η Αίγυπτος συμμετέχει οικονομικά πέρα από την ιδιοκτησία περίπου με το 1 τρίτο της συνολικής χρηματοδοτήσεως. Δεύτερο παράδειγμα, ανανεώσιμη, βασικό πρόγραμμα για ανανεώσιμη ενέργεια είναι κάτι διαφορετικό, δεν είναι πρόγραμμα, μελέτη είναι, σχέδιο ε, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κυρίως, έχουμε αναμειχθεί σε αυτό και στην Αίγυπτο βλέπουμε ότι πάνω από 10% χρόνο αυξάνεται η ανάγκη σε ενέργεια, αύξηση του πληθυσμού και η οικονομική ανάπτυξη οδηγούν σε αυτή την αύξηση κατανάλωση και πρέπει να αντιμετωπιστεί. Λοιπόν, έχει ορυκτούς πόρους, καύσιμα, φυσικό αέριο, Αίγυπτος. Αυτοί οι πόροι εξαντλούνται σιγά σιγά. Απ' την άλλη, η Αίγυπτος έχει ουσιαστικό δυναμικό για ηλιακή ενέργεια και αιωλική ενέργεια. Έχει δυνατότητες. Λοιπόν, σε αυτό το μέσο έχουμε το βασικό μας αρχικό σχέδιο. Θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο για την ηλιακή ενέργεια και να προετοιμάσουμε μελέτη σκοπιμότητας για την πρώτη κατάσταση ηλιακής ενέργειας στην Αίγυπτο. Η οικονομική συμμετοχή της, Ευρω... της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι 3 εκατομμύρια ευρώ και εμείς η KFW συνοδεύουμε τη μελέτη καταρχήν και προβλέπεται σε μεταγενέστερο στάδιο να χρηματοδοτήσουμε την πρώτη αυτή ηλιακή εγκατάσταση μονάδα παραγωγή ενέργεια μαζί με του εταίρου μα που χρηματοδοτούν και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τέλο, κάτι εξίσου σημαντικό. Αυτό συνάδει με το γενικό στόχο τη Ευρωπαϊκή Ενώση, του στόχου τη μάλλον, όσον αφορά την ηλιακή ενέργεια στη Μεσόγειο και η μελέτη θα είναι καταλήτη για μεταρρύθμιση του τομέα στην Αίγυπτο. Υπάρχουν κάποιες ανισορροπίες εκεί και θέλουμε να προωθήσουμε περιφερειακή και υποπεριφερειακή ενεργειακή συνεργασία μεταξύ χωρών. Τέλος, τελευταίο παράδειγμα, καταπίστευμα για την υποσαχάρια ε, Αφρική για ανάπτυξη Εκεί για τα ύδατα, στην Καμπάλα, για τα ύδατα και για τα υγρά απόβλητα, εκεί ο πληθυσμός δεν έχει σύστημα αποχαιρετευτικό. Δεν έχει πρόσβαση. Και στην πρωτεύουσα πολλά σημεία δεν έχουν καθαρό πόσιμο νερό. Το πρόγραμμα αυτό λοιπόν δημιουργήθηκε για να επεκταθεί η κατεργασία του ύδατος, η δυνατότητα διανομής του ύδατος και να βελτιωθούν οι υπηρεσίες, κυρίως και σε πρώην ε, κατοικημένες περιοχές, αν θέλετε. AFD ε και ERB ε έχουν χρηματοδοτήσει και η ITF ε και η FW έχουν συμβάλει. Όχι με δάνειο, αλλά με χορηγία στη συγκεκριμένη περίπτωση. Ποια είναι όλη εμπειρία μας. Πρακτικά τι είδαμε, τι διαπιστώσαμε όσον αφορά τον σχεδιασμό. Ο σχεδιασμός λοιπόν αυτός δημιουργεί ευνοϊκό παράδει, ε, περιβάλλον για καινοτόμες προσεγγίσεις και καλά προγράμματα και υπάρχει και ανταγωνισμός ιδεών. Τι εννοώ με αυτό. Είναι ένα πολύ ευέλικτο εργαλείο αυτό που χρησιμοποιούμε, πολύ ελκυστικό για χρηματοπιστωτικούς φορείς να έχουν πρόσβαση σε αυτούς τους πόρους οι χρηματοδοτιστικοί φορείς θέλουν να προσφέρουν αρκετά προγράμματα για να ανταγωνιστούν για τους πόρους που διατίθενται και η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να κάνει την επιλογή των προγραμμάτων εκείνων που ταιριάζουν με τους στόχους της. Δεύτερον, διευρύνει η αναπτυξιακή συνέπεια, αντίκτυπο που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και η ορατότητα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Διότι όλα αυτά που σα ανέφερα θεωρούνται σαν ευρωπαϊκή συνεισφορά σε ένα πρόγραμμα στο Μαρόκο, σαν ε, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και άλλους δωρητές, την Παγκόσμια Τράπεζα Φερρυπίν, με το Ταμείο της για την Καθαρή Τεχνολογία. Βελτιώνει την αποτελεσματικότητα της ενίσχυσης και δραματικά, αν δείτε τα προγράμματα που έχουμε προγραμματίσει για το Ίδωρ και λοιπά και για την ε, αυτοεξυπηρέτηση, να μπορούν να σταθούν οι ντόπιε αρχές στα πόδια τους, έχουμε μια, το κάνουμε αυτό έχοντας μια αιγίδα ευρωπαϊκή στη χρηματοδότηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θέλουμε να εκμεταλλευτούμε τις ιδέες των χρηματοδοτικών φορέων στους διαφόρους τομείς για να βρούμε συγκριτικά ωφέλη στους διάφορους τομείς που θέλουμε να καλύψουμε. Γίνεται επιμερισμός έργου μεταξύ χρηματοδοτικών οργανισμών, άρα υπάρχει ευελιξία, μπορούμε να θέτουμε καθήκοντα με ευελιξία και τέλος, εξίσου σημαντικό, μειώνεται το κόστος συναλλαγών. Οι εταίροι μας έχουν ένα χρηματοπιστωτικό οργανισμό ε, που πρέπει να φροντίσουν και να έρθουν σε επαφή με αυτόν. Λοιπόν, είμαστε σε θέση με αυτό το μέσο σχεδιασμού να χρηματοδοτούμε κατά περίπτωση, ε, διότι μπορούμε να ετοιμάσουμε πακέτα χρηματοδοτικά για κάθε περίπτωση λαμβάνοντας υπόψη το χρηματοδοτικό ε, δυναμικό των εταίρων μας και είμαστε σε θέση μέσω των πακέτων χρηματοδότηση μέσω πολλών δωρητών να χρηματοδοτήσουμε προγράμματα μεγάλη κλίμακα όπω στην Αίγυπτο, που είμαστε σε θέση εκεί να επηρεάσουμε σημαντικά μετατροπή του τομέα, μεταρρύθμιση, δημιουργούν κατάλληλο πλαίσιο και περιβάλλον που επιτρέπει την επιτυχία των διαφόρων προγραμμάτων και έργων στο τέλος της περίοδου. Ευχαριστώ. Και τώρα το λόγο η κυρία Μαλίνα Γκαλάρ. Good afternoon and thanks very much for inviting us to share our... Παρακαλούμε, ακούτε καλά η ελληνική διερμηνία. Μας λέτε αν ακούτε καλά την ελληνική διερμηνία, σας παρακαλούμε. Είμαστε διαθεσή σας. Ένα νεύμα σας παρακαλούμε. Blended funds from a number of IFIs and DFIs. And we would like to share with you some of the... Το κρίσιμο σημείο για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε αυτό, σε αυτό το σημαντικό θέμα. Όπως είπε και ο εισηγητής, φαίνεται να υπάρχει συνένεση μεταξύ των ευρωπαϊκών οργανισμών ότι χρειαζόμαστε πιο συνδυασμένα μέσα, αλλά πρέπει να ρωτήσουμε όντως μπορούμε να το προωθήσουμε. Για να διευκρινίσω λοιπόν αυτό το οποίο έχει περιπλέξει το θέμα, ε, μπορεί κανείς να συνδυάσει ε, τους, ε, τα δάνεια και τις χορηγίες σε διάφορα επίπεδα. Πρόκειται δηλαδή για δύο διαφορετικά στοιχεία τα οποία μέχρι στιγμής ενδεχομένως δεν είχαν κατανοηθεί σωστά. Η ερώτηση είναι χρειάζεται μεγαλύτερο μείγμα ή πόσο περισσότερο πρέπει να τα αναμίξουμε. Δηλαδή πρέπει να χρησιμοποιήσουμε χρησιμοποιήσουμε ε, τα, τους διαθέσιμους πόρους και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι χρειαζόμαστε μία τέτοια προσπάθεια και αυτό έχει γίνει με τα ε, concessional loans του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου το 2009. Όταν πρόκειται ε, για χρηματοδότηση από τον ιδιωτικό τομέα, όπου υπάρχει κάποια βοήθεια, όχι όμως ολόκληρη, αυξάνουμε επίσης. Αυξάνουμε και τις ε, πολυμερείς ε, ενισχύσεις. Είναι γενικές τάσεις αυτές οι μαύρες γραμμές για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε τον ιδιωτικό τομέα την τελευταία δεκαετία. Κατόπιν αυτού θα πρέπει στα πλαίσια αυτά να δούμε εφόσον υπάρχουν όλο και λιγότερες ε, χορηγίες από την Ευρωπαϊκή Ένωση που μπορούν να χρησιμοποιηθούν καλύτερα για να δούμε ε, ποιες ε, είναι οι διάφορες δυνατότητες και να λάβουμε μία απόφαση σύμφωνα με αυτό. Διότι λέτε στην έκθεση την οποία κάνετε για το Κοινοβούλιο ότι η πολυμερής βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ενώσεως είναι είναι προστιθέμενη αξία. Αυτό σημαίνει ε, συγχρόνως ότι πρέπει να πηγαίνουμε αντίθετη προς τους κύκλους, αντίθετα ε, ε, μην ακολουθούμε τις τάσεις της αγοράς και ό,τι έχει γίνει στο παρελθόν, αλλά να προσπαθήσουμε να χρησιμοποιήσουμε τα μέσα τα οποία έχουν έλλειψη. Τουλάχιστον όσον αφορά τις ευρωπαϊκές ε, ε, προσπάθειες και θα πρέπει να απαντήσουμε στο εξής ερώτημα. Ποιοι θεσμοί και ε, ποιοι οργανισμοί μπορούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να προσφέρουν αυτές τις προϋποθέσεις, διότι υπάρχουν δανειακές δανειακοί οργανισμοί από διάφορες πλευρές και ίσως οι δυνατότητες ε, που μπορούν να συγχρηματοδοτηθούν από την OIB ε, ε, δεν είναι πιο αποτελεσματική για την βοήθεια αυτή. Για ποιο λόγο, διότι υπάρχει ελάχιστη εμπειρία και επίσης διότι ε, το ο χρηματοοικονομικό μέσον στρέφεται ως επιτοπλίστων προς τη χρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα. Πρόκειται δηλαδή για τα κεφάλαια τα οποία απευθύνονται περισσότερο προς τον ιδιωτικό τομέα. Στις χώρες αποδέκτες το 70% των, της χρηματοδότησης αυτής απευθύνεται στον ε, ιδιωτικό τομέα και μόνο 30% στο δημόσιο και όπως σας είπα δεν πρέπει να ακολουθούμε μόνο την τάση της αγοράς διότι είναι πολύ πολύ σημαντική η ε, χρηματοδότηση του δημόσιου τομέα στις χώρες αυτές. Όταν λοιπόν απαντήσουμε στο πρώτο ερώτημα ε, του πόσο μπορούμε καλύτερα να χρηματοδοτήσουμε και ε, πόσο θα αναμίξουμε τα κεφάλαια, πρέπει να δούμε πώς η βοήθεια πρέπει να απευθυνθεί στον ιδιωτικό τομέα. Διότι μπορεί να υπάρξει χρηματοδότηση του ιδιωτικού ταμεία χωρίς ε, κεφάλαια ενισχύσεων. Η Παγκόσμια Τράπεζα ε, κάνει αυτού του είδους τις επιχειρήσεις ε, για το μακρύτερο χρονικό διάστημα. Μας λέγουν όμως δεν μας αρέσει ε, η ευρωπαϊκή ενίσχυση να βοηθά τις ε, χώρες με χαμηλό εισόδημα διότι καταστρέφει την αγορά. Δεν θέλω να σας πω ότι εγώ συμφωνώ με αυτή την άποψη αλλά σας λέω ότι έχουμε δει στις περιπτώσεις αυτής. Και αυτό το οποίο μπορούμε να πούμε σε αυτό το είδος δανεισμού για το 70% των ε, επενδυτικών ε, ταμείων για τις χώρες ΑΚΕ είναι ότι δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι είναι πολύ αποτελεσματικές και εδώ διαφωνώ με τους Άγγλους ομιλητές δεν θα επισέλθω σε λεπτομέρειες ε, κάναμε όμως μία μελέτη και θα σας αφήσω μετά κοντά στην είσοδο αντίγραφα για τα προγράμματα τα οποία έχει χρηματοδοτήσει η IFC η οποία βοηθάει τον ιδιωτικό τομέα και ε, έχουμε εντοπίσει διάφορα προβλήματα. Καταρχήν, δεν ξέρουμε πώς ε, ο δανεισμός αυτός ε, συνάδει και κατά πόσον συνάδει με ε, την αρχή της ε, αποτελεσματικότητας σε σχέση με το κόστος. Επίσης, η απόδοσή τους δεν είναι τόσο καλή. Ε, δεν έχω τώρα χρόνο να επισέλθω σε λεπτομέρειες, σε συνέχεια ευχαρίστως. Επίσης, όσον αφορά το χαρτοφυλάκιο των, των εταιριών αυτών, και της χρηματοδοτήσεως αυτές ε, πηγαίνει στις μεγαλύτερες εταιρείες. όταν δείτε ποιες εταιρείες χρηματοδοτούνται βλέπουμε ότι είναι στρεβλωμένη η κατάσταση και αυτές ε, είναι οι διαπιστώσεις τις οποίες έχουμε κάνει και βλέπετε ε, ποιος χρησιμοποιεί τη χρηματοδότηση από αυτόν τον οργανισμό. Βλέπουμε λοιπόν ότι ιδίω χρηματοδοτούνται οι πολυεθνικές εταιρείες ε, του ΟΣΑ. Και ένας από τους μηχανισμούς που έχει χρησιμοποιηθεί μέχρι στιγμής για να διοχετεύσουμε τη χρηματοδότηση αυτή σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις στις χώρες αυτές οι οποίες χρειάζονται περισσότερες πιστώσεις, πολύ περισσότερο από τις πολυεθνικές εταιρείες ε, είναι χρηματοοικονομικοί μεσάζοντες οι οποίοι αυτή τη στιγμή χρησιμοποιούνται από την ε, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεως και βλέπουμε ότι δεν είναι ο καλύτερος τρόπος για να υπάρξουν αποτελέσματα. Παραδείγματο χάρη είναι εταιρείε ε, ε, private equity και δεν ε, μπορούμε να δούμε πώς αυτές, αυτοί οι οργανισμοί όντως μπορεί να αποδώσουν. Πρέπει λοιπόν να δούμε αν το νέο αυτό σχήμα θα ασχοληθεί με, το ίδιο, με την ίδια μορφή. Και τέλος, η Ευρωπαϊκή ε, Τράπεζα ε, ε, Επενδύσεως και οι περισσότερες από αυτές τις εταιρείες βρίσκονται εγκατεστημένες σε φορολογικούς παράδεισους. Πράγμα το οποίο δείχνει ότι ε, έτσι διοχετεύονται τα χρήματα ε, προς τις χώρες αυτές και θα πρέπει σε το επόμενο πολιετές ε, πρόγραμμα να δούμε τι χρήματα θα οδεύσουν προς αυτές τις εταιρείες και να διαπιστώσουμε το εξής. Να δούμε πολύ προσεκτικά και να σκεφτούμε τι χρήματα πρέπει να στέλνουμε εις τον ιδιωτικό τομέα. Τι χρειάζεται τι, ε, ε, τι μηχανισμοί χρειάζονται και ίσως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να μας βοηθήσει σε αυτή τη διαπίστωση. Δεύτερον, ε, εφόσον θα κοιτάξουμε τις διάφορες οργανώσεις και πώς αυτές κινούνται και πώς έχουν επιτύχει πιο αποτελεσματικά επιδόσεις, θα δούμε ότι ε, στο επόμενο πρόγραμμα θα πρέπει να προβλέψουμε ότι ε, θα χρειαστούν διάφοροι μηχανισμοί προστατευτικοί, θα πρέπει ε, να υπάρχουν διάφορα συστήματα τα οποία θα υπάρχουν θα ε, ε, υπάρξουν πολιτικές οι οποίες θα εξασφαλίζουν ότι περισσότερη χρηματοδότηση θα πηγαίνουν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αντί για τις πολυεθνικές και όπως είπε και ο προλαλής σας, ε, δεν έχει σταματήσει αυτή η ενίσχυση αλλά βλέπετε τα αποτελέσματα δεν είναι λαμπρά. Τέλος, τι προσπαθούμε να επιτύχουμε ε, πρέπει να υπάρξει επιπλέον και έλεγχος για να δούμε ότι ε, καμία χώρα η οποία, ή καμία εταιρεία η οποία βοηθείται με αυτόν τον τρόπο δεν προέρχεται από φορολογικούς ε, παραδείσους. Δίνω τώρα το λόγο στον κύριο Γκέρχαρτ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Thank you, Madam Chair. Honourable Members of Parliament, ladies and gentlemen. Κυρίες και κύριοι, σας ε, ευχαριστώ που μου επιτρέπετε να μιλήσω σήμερα και ε, θα κάνω μία παρουσίαση. And some factual data, if I can find it here. I think it's it. Θα προσπαθήσω να σας παρουσιάσω διάφορα στοιχεία τα οποία ψάχνω αυτή τη στιγμή. minute for me, um, Χίλετ, υπεύθυνο των ε, θεμάτων υποδομών στην ε, ΤΕΦΚΟ και θα ήθελα να σας μιλήσω για το θέμα αυτό από τότε που η ομάδα εργασίας έκανε την αναφορά στο Συμβούλιο του 2009 και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουμε διάφορα ε, μέσα ενεργά εδώ και μέσα για θέματα ψυχικής βοήθειας. Θα σας δώσω κάποια στοιχεία. Δεν θα σας δεν θα μακρηγορήσω παρουσιάζει τι λεπτομέρειες, την έχετε στη διαθεσή σα Θα προσπαθήσω να επικεντρωθώ στις αρχές του συνδυασμού και των επιπτώσεων της πράσινης βίβλου. Είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε ότι για τον συνδυασμό που χρησιμοποιείται ασχολούμεθα κυρίως το συνδυασμό των ε, ε, υποδομών σε θέματα μεταφορών ενέργειας. Θέλουμε να υποστηρίξουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι τομείς που καλύπτονται είναι η μεταφορά, η ενέργεια, οι νέες τεχνολογίες, οι κλιματικές αλλαγές, θέματα περιβάλλοντος, θέματα υγείας, παιδείας, υποστήριξη του ιδιωτικού τομέα και κυρίως εστιάζει προσπάθειές μας στις χώρες τις οποίες στον ε, τομέα της θέλησης και της εκπαίδευσης υπάρχουν μεγάλα προβλήματα χρηματοδότησης, δηλαδή χρησιμοποιούνται στους τομείς αυτής ε, δάνεια και χορηγήσεις προς τις χώρες τις πιο φτωχέ που είναι την περισσότερη ανάγκη. Όπως σας είπα, οι κύριε αρχέ είναι ότι η αναπτυξιακή μας πολιτική είναι ο κύριος, η κύρια κινητήρια δύναμή μας, δηλαδή εστιαζόμαστε σε μία ε, πολιτική συμπερίληψη όνων, με αυτού του συνδυασμένου μηχανισμού προσπαθούμε να προωθήσουμε του προτεραιότητε τι οποίε έχουμε στον αναψηφιακό τομέα κάνοντας συμπληρωματικές ενέργειες με τις στρατηγικές περιφερειακής και εθνικής πολιτικής. Πρόκειται για ένα μέσον λοιπόν συμπληρωματικό σε σχέση με αυτά τα οποία υπάρχουν και με τα περιφερειακά ή τα άλλα εθνικά αναπτυξιακά προγράμματα. Η δυνατότητα χρηματοδότησης ε, σε νέα κονδύλια το ε, επιτρέπει με δανεισμό και άλλων εταίρων με άμεσες ε, επενδύσεις εκ μέρους άλλων και ελπίζουμε ότι με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουμε να προσελκύσουμε και κονδύλια και πιστοτικά ιδρύματα του ιδιωτικού τομέα σε τομείς ε, τις οποίους δεν θα μπορούσαν με να στοχεύσουμε σε διάφορες χώρες διαφορετικά. Επίσης, υπάρχει προσπάθεια αηφορίας και αυτό το οποίο μας ε, απασχολεί κυρίως είναι η αηφόρος ανάπτυξη. Όλα αυτά γίνονται στα πλαίσια του άρθρου 4 των διαβουλεύσεων με το FMI. Θέλουμε να έχουμε ε, διάλογο με αυτούς οι οποίοι θα μας βοηθήσουν να έχουμε συνδυασμό δανείων και χορηγήσεων και αηφόρο δανεισμό. Τώρα, όσον αφορά τα διάφορα προγράμματα, θέλουμε να είναι υγεία από τεχνικής και χρηματοδοτικής άποψης. Πρέπει να γίνουν στην αρχή μελέτες κοπιμότητας για να δούμε κατά πόσον τα πακέτα τα οποία χορηγούμε ε, αρμόζουν. Θέλουμε οι συνθήκες αηφορίας να ισχύουν ακόμη και μέχρι να ολοκληρωθούν τα διάφορα project και κυρίως μετά και θέλουμε κίνητρα ώστε να μπορούν να δίδονται και διάφορα ε, άμεσα δάνεια και χορηγήσεις. μείωση του κινδύνου, αξιολόγηση που αποτελεί μέρος του προγράμματος, μελέτη αξιολόγησης κινδύνων, αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα της ε, κρατικών προμηθειών και εφαρμογή και ε, επιτήρηση της όλης εφαρμογής των σχεδίων. Ποια είναι η προστιθέμενη αξία αυτών των συνδυασμών. Η μόχλευση η δυνατότητα της Επιτροπής να συμμετέχει στην χρηματοδότηση μεγαλύτερης εμβέλειας έργων υποδομής, συμμετοχή και με άλλες χρηματοδοτικές ε, ε, οντότικες, εφαρμογή ε, των συντονιστικών μέτρων εκ μέρους όλων των δωρητών, εναρμόνιση των διαδικασιών σύμφωνα με την ατζέντα Άκρα και Παρισιού. Όλα αυτά στα πλαίσια των ρυθμίσεων που λαμβάνουμε, ώστε να μπορεί η ορατότητα όλων αυτών των ε, σχεδίων συνδυασμού και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κομισιόν ιδιαίτερα να αυξηθεί. Πιστεύουμε ότι όλα αυτά γίνονται ε, σύμφωνα με την διακήρυξη του Παρισίου. Χρησιμοποιούμε το σύστημα των ε, ε, δικαιούχων κρατών. Θέλουμε να θέσουμε όλοι από κοινού τα κονδύλια τα οποία διαθέτουμε. Θέλουμε να είμαστε υπεύθυνοι για όλες αυτές τις διαδικασίες, να μπορούμε να ασκούμε και τον συντονισμό όλων των Ευρωπαίων δωρητών. Ε, όλα αυτά βεβαίως ε, στα πλαίσια της ε, πρόθεσης του διαλόγου ώστε να υπάρχει πολύ καλή οικονομική δίκηση και διαφάνεια σε όλες αυτές τις διαδικασίες. Μέχρι τώρα ποια είναι τα αποτελέσματα αυτών των κυρίων σχεδίσεων. Ε, το EU Africa Infrastructure Trust Fund από το 2007 έχουν χρησιμοποιηθεί στα πλαίσια αυτής της συνεργασίας, ε, έχουν εγκριθεί στα πλαίσια της συνεργασίας 35 διαφορετικά σχέδια, έχουν εγκριθεί κονδύλια 240 εκατομμυρίων και υπάρχει και το δεύτερο σχέδιο ε, για την σχέδια επενδύσεων γειτονίας με την ε, βόρεια, χώρες της Βόρειου και Νοτιού Μεσογείου, όπου έχουμε 39 σχέδια και 275 εκατομμύρια τα οποία έχουν εγγύθει. Όλες τις συμπροματικές πληροφορίες τις έχετε εδώ στις σχετικές ε, ιστοσελίδες που βλέπετε στην οθόνη. Μου ζητήθηκε να πω και κάποια λόγια για την το βήμα αυτό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για την σχέση του με την Πράσινη Βίβλο. Δεν έχω προετοιμάσει γραπτός τίποτε για αυτό το θέμα. Όσον αφορά αυτή την EU πλατφόρμα, οι συζητήσεις δηλαδή μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων, ο διάλογος συνεχίζεται. Η ομάδα εργασίας θα θέσει τους όρους για να μπορέσει να υπάρξει διάλογος, η εντολή έχει συζητηθεί και συμπεριλαμβάνονται αρχές εναρμόνισης του συνδυασμού των μέσων που εφαρμόζονται βάσει των ε, για να δούνε πώς θα αξιολογηθούν τα κριτήρια που θα ε, πρέπει να πληρούνται και πώς θα χρησιμοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ο συνδυασμός αυτής της χρηματοδότησης. Η Επιτροπή λέει ότι η συμμετοχή των κρατών μελών θα πρέπει να είναι ελεύθερη και ανοιχτή, καθώς και η συμμετοχή ενδεχομένων των ε, χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως της Ευρωπαϊκής Τράπεζας. Ακόμη δεν έχουν ολοκληρωθεί όλες οι διαδικασίες. Ίσως ο συνάδελφος Άλεξ Τζόνς θα μπορούσε να προσθέσει κάτι. Τίποτε όμως ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί. Ο σχεδιασμός δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ως η εναλλακτική λύση, θα πρέπει να συνδυαστεί και με διάλογο και να δούμε πώς θα μπορέσουν σε ευάλωτες οικονομίες με μικρά εισοδήματα και σε χώρες ε, που έχουν δύσκολη οικονομική κατάσταση να γίνουν αποδεκτά τα σχέδια τα οποία θέλουμε να ε, εφαρμόσουμε. Όλα αυτά βεβαίως θα πρέπει να έχουν κατά κύριο στόχο την αναπτυξιακή πολιτική σύμφωνα με τα συμπεράσματα στα οποία καταλήγει η πράσινη βίβλος. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να γίνει από αυτόν τον πολιτικό διάλογο, στον οποίο να συμμετάσχουν ο δημόσιος και ο ιδιωτικός τομέας που θα κληθούν να χρηματοδοτήσουν πράξεις και ενέργειες για να υλοποιηθούν οι στόχοι αυτής της πολιτικής. Η ιδέα να χρησιμοποιηθούν τα υπάρχοντα μέσα στο πλαίσιο του δυνατού και να έχουμε ε, περισσότερες ε, χρηματοδοτήσεις εκ μέρους των χρηματοπιστωτικών ε, ιδρυμάτων είναι από τους στόχους μας. Ευχαριστώ, σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η κυρία Κρήτου έχει το λόγο. Thank you very much, Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Καταρχάς, να ευχαριστήσω τον κύριο Κάσμαρεκ, τον συνεισηγητή, και να τον συγχαρώ για την έκθεση Συνάμα. Θα ήθελα επίσης να τον ευχαριστήσω για την πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Τίθεται πολλά θέματα. Κοινωνικά, περιβολαντικά. Έχω όμως κάποια σχόλια και προτάσεις. Πρώτα απ' όλα, χρειάζεται αυξανόμενος μεγαλύτερος ρόλος για την ανάπτυξη στο δημοσιονομικό αυτό το πολιτες πλαίσιο. αναθεωρήθηκε πολλές φορές από όταν εγκρίθηκε το 2006. Κάτι άλλο που λείπει, σημαντικό, το 0,7% του ΑΕΠ να διατίθεται για την επίτευξη των στόχων της χιλιετίας με καλύτερο έλεγχο και συνεκτική πολιτική για ανάπτυξη. Δύσκολο να υποχρεώσει τα κράτη-μέλη να το κάνουν αυτό. Να τηρήσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις και καθήκοντα τώρα την περίοδο της κρίσης. Και είναι σημαντικό να αναφέρεται ρητά ότι παροτρύνουμε τα κράτη-μέλη να τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους. Και η οικονομική ανάπτυξη πράγματι μπορεί να είναι κινητήρα σημαντικό για την ανάπτυξη, το υποστηρίζω. Μπορεί α, μόνο αν μειωθούν οι ανισότητες να εκριζώσει την φτώχεια, που είναι ένα πρόβλημα στις αναπτυσσόμενες χώρες. Στην Επιτροπή Γυναικών, κατόπιν πρωτοβουλία μου, πρότεινα τροπολογίες για τη συμπερίληψη του θέματος της των φύλων που έλειπε από την έκθεση. Και το ψήφισε την περασμένη εβδομάδα η Επιτροπή Γυναικών. Η ισότητα των γυναικών και η ενίσχυση και υποστήριξη των γυναικών στα οικονομικά και πολιτικά θέματα και τα ανθρώπινά του δικαιώματα είναι ουσιαστικά για βιώσιμη ανάπτυξη και μείωση τη φτώχεια. Όταν μιλάμε για ενίσχυση, θα πρέπει να σκεφτόμαστε τι γυναίκε, τα παιδιά και, του ανθρώπου με αναπηρίες. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ντέβα έχει το λόγο. Εκ μέρους τους, της συναδέλφου της κυρίας Μακλόχλιν, που είναι σκιώδης εισηγήτρια στην ομάδα μου και δυστυχώς δεν μπορεί να παραστεί, θέλω να πω κάποια από τα σχόλια που είχε. Θεωρεί ότι αυτή η δουλειά μπορεί να έχει μεγάλες συνέπειες και να επιφέρει συνολική ανάπτυξη και ανάπτυξη ιδιωτικού τομέα, που είναι σημαντικό για την αναπτυξιακή πολιτική. Τώρα, το πώ οι φορεί του ιδιωτικού τομέα μπορούν να βοηθήσουν καλύτερα το δημόσιο τομέα είναι κάτι πολύ σημαντικό και να εστιαστούν εκεί οι προσπάθειε. Είχαμε το θέμα των μικροπιστώσεων και μικροχρηματοδότηση. Είδαμε ότι υποστηρίζουν κατά πολύ την ανάπτυξη. Έχουν τεράστιε συνέπειε. Τα προγράμματα αυτά πρέπει να είναι διαφανή και ελεγχόμενα. Η ασφάλεια του νερού, το θέμα του νερού, είναι πολύ ζωτική σημασία για την ανάπτυξη. Εντυπωσιάστηκα από τα στοιχεία. Ο τομέα των υδάτων υπογραμμίστηκε στα αυτά τα μεικτά προγράμματα των εταίρων μα για αναπτυξιακά ζητήματα. Εντυπωσιάστηκα τα μάλα με αυτά που υπόθηκαν μέχρι τώρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Σαρτζεντίνη έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον κύριο Κασμάρεκ για την γνωμοδότησή του καθώς επίξει και τους ο, τρεις ε, τρεις εμπειρογνώμονες που μας μίλησαν για blending. Ήξερα τι, το νόημα, αλλά δεν είχα ακούσει ε, αυτή την ε, νέα ιδέα. Θέλω να θέσω ένα ερώτημα που θεωρώ ότι είναι πολύ ουσιαστικό. Γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ε, ξεκινήσει τώρα μία πράσινη βίβλο για να αναθεωρήσει την αναπτυξιακή ανθρωπιστική βοήθεια στα μέσα μιας οικονομικής κρίσεως. Δεν επηρεάζεται η αποτελεσματικότητα, οι ανάγκες που μπορεί να οδηγήσουν σε επιχειρήματα σύμφωνα με τα οποία μπορούμε να πούμε ότι με λιγότερα χρήματα μπορούμε να επιτύχουμε τα ίδια ίσως και περισσότερα. Το ίδιο ισχύει και στην ιδέα του blending ε, του, του μείγματος. Ε, αν ε, συνδυάσουμε διάφορες μοτέφες χρηματοδοτήσεως θα έχουμε περισσότερα αποτελέσματα με λιγότερα χρήματα. Εγώ αμφιβητώ. Θα υπάρχει διαφάνεια. Θα βλέπουμε τι είναι τα αποτελεσματικότητα των, τα αποτελέσματα αυτών των χρημάτων. Ε, μετά ε, μία ερώτηση στον κύριο Κάσμαρεκ, τον εισηγητή και στην αδερφό μου, αλλά και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τι είναι αυτή η μορφή αναπτύξεως την οποία πρεσβεύεται. Εγώ θα ήθελα να ξέρω ποιο είναι το νόημα αυτής της ανάπτυξης μετά από την ε, συμφωνία μας σχετικά με την ανάπτυξη διότι μιλάμε για ανεπαρκή ανάπτυξη εδώ και πολύ καιρό. Θυμάμαι ότι την πρώτη φορά που προσπάθησα να ε, προφέρω αυτές τις λέξεις ε, αναρωτιόμουν τι είναι. Τώρα όμως μιλάμε για poor growth αντί για inclusive growth. Και τι εννοείται, τι εννοείται ακριβώς. Εάν λοιπόν θυμόμαστε ότι πολλές χώρες ε, και εξετάζουν το ποσοστό της του OBA. Εμείς ε, μειώσαμε το 0,8 στο 0,7, οπότε τι είναι το ODA, ποιος είναι ο ορισμός του. Έχει δοκιμαστεί και στο παρελθόν, θα το ξαναδοκιμάσουμε και τώρα. Θεωρώ ότι δεν είναι κατάλληλη στιγμή να προσπαθήσουμε να διατυπώσουμε νέες αναπτυξιακές ιδέες σαν τρόπο να δικαιολογήσουμε γιατί μειώνουμε τις ε, δαπάνες μας και τις επενδύσεις μου. Ε, αυτά είναι προς το παρόν. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μαρτίνες έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να τονίσω πόσο εξαιρετική είναι η έκθεση του φίλου μου κυρίου Κασμάρεκ και θα ήθελα κυρίως να τονίσω το εξής. Οι διερμηνεί ζητούν στον κύριο Μαρτίνες να μιλάει στο μικρόφωνο ή τον ακούνε. Επαναλαμβάνει ο κύριος Μαρτίνεφ. Μου φαίνεται εξαιρετική η έκθεση του συναδέλφου Κασμάρεκ. Πρόκειται για λογική ισοσκελισμένη έκθεση και θα ήθελα κυρίως να τονίσω ότι στην έκθεση αυτή υπάρχει κάτι το οποίο συζητήσαμε σήμερα το πρωί όταν μιλήσαμε για την έκθεση του κυρίου Γκέριντ. Δηλαδή, κάτι το οποίο λείπει στα περισσότερα έγγραφα παρά το γεγονό ότι αυτό το θέμα αναφέρεται μόνο στις παραγράφους 22 και 23. Πρόκειται για την ε, επιστηστική ασφάλεια και την γεωργία, την ασφάλεια των ε, ειδών διατροφή. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να τονίσουμε τώρα που βλέπουμε πώς εξελίσσονται τα πράγματα ανά το κόσμο και αν ε, δούμε τι συμβαίνει στα πλαίσια της Συμφωνίας Κοτονού. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να γίνει εκ μέρους όλων των χωρών προσπάθεια για να δοθεί προτεραιότητα στο θέμα αυτό της εξασφάλισης της ε, ασφάλειας των ειδών διατροφής. Και συγχρόνως να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε μια γεωργία την οποία πολλές φορές αφήνουμε κατά μέρο στις αναπτυσσόμενες χώρες, όπως και στις, συνέβη δικές μας χώρες. Δηλαδή, τα άτομα τα οποία ασχολούνταν με τη γεωργία πολλές φορές τα ξεχνάμε και δεν ακολουθούν την ίδια οικονομική ανάπτυξη που υπάρχει και σε άλλους τομείς. Εν πάση περιπτώσει, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον φίλο μας, τον κύριο Κασμάρεκ, ο οποίος στις δύο τελευταίες παραγράφους της έκθεσής του το ανέφερε αυτό το θέμα. Επίσης θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο το οποίο δεν έχει μεγάλη σχέση με το θέμα μας, αλλά είναι και αυτό επίκαιρο. Πρέπει να πω το εξής, αγαπητοί συνάδελφοι. Όλο και περισσότερο πρέπει να πω ότι εξοργίζομαι. Είμαι παραξενεύει το ότι κάθε φορά που έχουμε μπροστά μας εμπειρογνώμονες, ακούμε να χρησιμοποιούν όρους τεχνικούς που δεν καταλαβαίνουμε καθόλου. Όλο και περισσότερο. Εκατομμύρια εκατομμύρια και εκατοντάδες όρους που είναι εκεί για τους εμπειρογνώμονες, αλλά για τους περισσότερους από μας είναι ακαταληπτή. Ίσως εμείς το 25% το καταλαβαίνουμε, αλλά ο κοινό συνητός 0% καταλαβαίνει. Και έτσι υπάρχει αυτή η μεγάλη απόσταση μεταξύ αυτών που μιλούν με τεχνική όρου και αυτών στου οποίου απευθύνεται που δεν καταλαβαίνουν τίποτε. Θα πρέπει λοιπόν διάφορες έννοιες πολύπλοκες που παρουσιάζονται και με κρυπτογραφικό τρόπο, εμείς τι να κάνουμε, να το καταπιούμε, να το χωνέψουμε για να το μεταφέρουμε και στον κοινό αφνητό. Τι να κάνουμε. Το λέγω αυτό διότι έχουμε δυσκολία με όλους αυτούς τους όρους. Πιστεύω ότι το πρόβλημα που έχουμε αυτή τη στιγμή, ένα από τα βασικά προβλήματα που έχουμε αυτή τη στιγμή, είναι το θέμα της επανακοινωνικοποίησης κάποιων διαδικασιών για να μπορέσουμε να κινητοποιήσουμε τους λαούς μας και στην Βόρεια και στην Νότια Ευρώπη. Και αν αρχίσουμε να τους μιλάμε ακατανόητα με όλες αυτούς τους ώρες, δεν θα μπορέσουμε ούτε να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο, ούτε να τον κινητοποιήσουμε. Και αν δεν το κάνουμε αυτό, να συνεχίσουμε να γυρίζουμε γύρω-γύρω όλοι, στη μέση ο Μανώλης και δεν θα κάνουμε καμία πρόοδο προς αυτό την κατεύθυνση που πιστεύω και δεν θα εμβαθύνουμε σε αυτά τα οποία συζητούμε και θέλουμε να κάνουμε, πράγμα το οποίο θεωρώ απαραίτητο. Θα ήθελα λοιπόν να πω ότι θα έπρεπε κάπως να μας διευκολύνουν κάποιοι με την κατανόηση των ε, ε κειμένων ε, και των παρουσιάσεων που μας γίνεται. Και θα πρέπει να πω το μεγάλο πλεονέκτημα της έκθεσης του κυρίου Κεσμάρκη είναι ότι είναι ευανάγνωστη από την πρώτη ως την τελευταία ε, λαστή φράση. Ούτε εκατομμύρια κρινήμοι υπάρχουν, ούτε κρυπτογραφημένοι όροι που μας μπερδεύουν. Και εφόσον εκπροσωπούμε τους πολίτες μας, θα πρέπει να κατανοούμε αυτά που μας λέγονται σε εμάς, να μπορέσουμε να τους εξηγήσουμε και σε εκείνους. Ευχαριστώ λοιπόν, ευχαριστώ και πάλι τον συνάδελφο για αυτά τα οποία είπε, τα οποία είναι χρήσιμα και αποδεικνύουν ότι έγινε εξαιρετική εργασία, αλλά θα ήθελα να ζητήσω και στους εμπειρογνώμονες που κάνουν πολύ καλή δουλειά να καταλάβουν ότι ώρες-ώρες απευθύνονται σε άτομα τα οποία δεν έχουν τον ίδιο κωδικό με αυτούς για να αποκρυπτογραφήσουν αυτά τα οποία μας ε, ε, λέγουν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ που με ακούσατε. Έχω δύο ερωτήσεις προς τους ειδικού σχετικά με αυτά που παρουσίασαν. Ένα ερώτημα αφορά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είπατε ότι φεύγετε να προσπαθείτε να αποφύγετε συνοστισμό. Πώς το κάνετε αυτό. Ποια μέτρα για να, αποφύγετε, να το αποφύγετε αυτό. Δύο-τρεις ανέφεραν το θέμα της ορατότητας της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, ότι με την ανάμιξη των πολιτικών αυτή τη μεικτή προσέγγιση θα βελτιωθεί, θα αυξηθεί με το blending. Πώς το επιτυγχάνει αυτό, αυτή η διαδικασία. Λοιπόν, θα δώσω το λόγο στους επαΐοντες για να απαντήσουν. Ο κύριος Ρόης ίσως μπορεί να εκπροσωπήσει τους εμπειρογνώμονες για να δώσει κάποιες απαντήσεις. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αυτή η ανάμειξη, αυτό το κράμα πώς βελτιώνει την ορατότητα. Το blending. Έδωσε ένα παράδειγμα στο Μαρόκο εγκατάσταση ηλιακή παραγωγής ενέργειας, ανανεώσιμε πηγέ ενέργειας. Με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης συνεργαζόμαστε. Ουσιαστική χρηματοδότηση γίνεται και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε και την Αφρικανική Ανεπτυξιακή Τράπεζα και την Παγκόσμια Τράπεζα με το Ταμείο τη για την ε, Καθαρή Ανάπτυξη. Άρα πολυσχηδέ μοντέλο. Και οι Ευρωπαίοι ομαδοποιούμαστε μαζί με τα ποσά που δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συνεργαζόμαστε για την υλοποίηση του προγράμματος. Μας βλέπουν εκεί. Δεν μας βλέπουν μόνο σαν KFW, σαν Ευρωπαϊκή Πτέρυγα, ένα consortium τραπεζών μας βλέπουν. Συν Ευρωπαϊκή Επιτροπή που διευθύνει το πρόγραμμα. Ε, πιστεύω ότι είναι πολύ καλό παράδειγμα αυτό που είπα. Άρα βελτιώνεται η ορατότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του το τρόπος. Για το δεύτερο ερώτημα και σε αυτό να απαντήσω. Για αυτό το crowding out. Πρέπει να κάνουμε διαφοροποίηση. Δεν συνεργαζόμαστε με ιδιωτικούς φορείς αν το δημόσιο τομέα. Στα πλαίσια των ε, διαφόρων επενδύσεων. Ο δημόσιος τομέας είναι ο εταίρος μας. και πώς βλέπουμε ω καλύπτει τις ανάγκες του τι κεφαλουχικέ ο δημόσιο τομέα για τα διάφορα έργα. Και αυτές οι χώρες μέσω εισοδήματος μόνο μέσω ιδιωτικών τραπεζών και κεφαλαγοράς μπορούν να πραγματοποιήσουν τους στόχους τους. Και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλύπτουμε τη διαφορά, τα κενά που έχουν στην προσπάθεια που κάνουν για να χρηματοδοτήσουν τα έργα τους. Οι άλλοι εμπειρογνώμονες έχουν κάτι να προσθέσουν, να σχολιάσουν, να ολοκληρώσουν τις απαντήσεις που δίδονται. Ωραία. Merci. Ευχαριστώ. Ναι. Ε, Είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς από το έγγραφο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως τι είναι η ευξημένη ορατότητα, διότι εμείς θέλουμε επίσης να εξαλείψουμε τη φτώχεια αλλά δεν έχω λάβει απάντηση. Για τον συνάδελφο από την Ισπανία θα ήθελα να πω τα εξής. Μετά την κρίση μάθαμε ότι η Ευρωπαϊκή οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις χρειάστηκαν να χρηματοδοτήσουν μαζικά τον ιδιωτικό τομέα επειδή δεν ήταν ρυθμισμένος. Ε, ε, νομίζω ότι εδώ είμαστε αντίθετοι στο ρεύμα, διότι έχουμε μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στις κεφαλαίες ιδίως στις χώρες με χαμηλό εισόδημα και θα προσπαθήσουμε να χρηματοδοτήσουμε τον ιδιωτικό τομέα, οπότε πιστεύω ότι όλοι πρέπει κάπως να προετοιμαστούμε για αυτά τα οποία έχουμε κατά νου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τους εμπειρογνώμενους οι οποίοι μας παρουσίασαν τα διάφορα θέματα και τώρα θα προχωρήσουμε στην εξέταση ε, της εκθέσεως του κυρίου Κασμάρεκ. Κυρία ε, κυρία ε, Πρόεδρε, και εγώ θα ήθελα να ακούσω τι έχει να πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οπότε, θα περιμένει ο κύριος Κασμάρεκ μέχρι να απαντήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. η αποφυγή του crowding out σημαίνει ότι το δίκτυό μας των αντιπροσωπιών Ευρωπαϊκής Ενώσεως θα μπορέσει να μας επιτρέψει να εντοπίσουμε ε, που ε, συμμετέχει περισσότερο ο ιδιωτικός τομέας από ό,τι παραδείγματο χάρη στην ε, ε, υποσαχάριο Αφρική και μετά θα κάνουμε διαβουλεύσεις με αυτές τις εκπροσωπήσεις μας για να δούμε τι προγράμματα μπορούν να προσελκύσουν κεφάλαια του ιδιωτικού τομέα και πιστεύω ότι κατά αυτόν τον τρόπο θα μπορέσει να υπάρξει μία συμμετοχή στις συζητήσεις και άλλων στοιχείων και αυτό γίνεται ε, σε συνεργασία με το δίκτυό μας και αναλόγως των εντοπίων συνθήκων. Αυτό είναι ο τρόπος με τον οποίο θα σας έλεγα ότι προσπαθούμε να αποφύγουμε το crowding out. Ο κύριος Κασμάρεκ έχει το λόγο τώρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε θα ήθελα να αναφέρω διάφορα σχόλια σχετικά με το blending και με άλλα θέματα που προέκυψαν κατά τη συζήτηση αυτή. Ευχαριστώ για τις παρουσιάσεις, παρόλο που και εγώ ε, είχα την ίδια εντύπωση. Δηλαδή, μετά τους εμπειρογνώμονες έχουμε περισσότερες ερωτήσεις παρά έχουμε λάβει ήδη απαντήσεις έχουμε περισσότερα ερωτηματικά. Αν όμως αυτό μπορεί να με βοηθήσει να καταρτήσω την έκθεσή μου, ε, θα το δεχτώ. Οι τροπολογίες από την Επιτροπή των Γυναικών είναι πολύ ουσιαστικές και τις ε, δέχομαι διότι το στοιχείο του mainstreaming της ισότητας των φύλων δηλαδή θα πρέπει να ισχύσει και μην ανησυχήσετε ε, θα αντικατοπτρίζονται στο τελικό κείμενο όλες οι ανησυχίες σχετικά με αυτό που ελέγχθη για ορισμένους κινδύνους. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι δεν μπορούμε να χαμηλώσουμε ε, το επίπεδο του ODA κατά 0,7 ε, το έχουμε ήδη πει, το λέμε εδώ και πολύ καιρό και κάθε φορά επαναλαμβάνουμε ότι εάν υπάρχει αλλαγή στην αναπτυξιακή πολιτική δεν πρέπει αυτό να γίνει εις βάρος της ε, βάσεως της αναπτυξιακής πολιτικής ε, που συζητείται στο επίπεδο ODA, δηλαδή 0,7. Αυτό το έχουμε αναλάβει κατά κόρον. Βεβαίως θα πρέπει ε, να ε, αναπτύξουμε ένα πιο πλούσιο μείγμα για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Ε, συγκεντρωτική ανάπτυξη. Συμφωνώ με αυτό που είπε η κυρία Σαρζεντίνη. Η απάντησή μας είναι συγκεκριμένη. Γνωρίζουμε τι εννοούμε όταν μιλάμε για συνολική ανάπτυξη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιτροπή συμφωνεί με ε, τον ορισμό μας. Η ανάπτυξη αυτή είναι μια ανάπτυξη που δεν αναφέρεται μόνο στον ενεργό πληθυσμό, όχι μόνο στα άτομα τα οποία μπορούν να δραστηριοποιηθούν, αλλά και ε, τα ε, παθητικά άτομα δηλαδή τα άτομα στα οποία θα καταλήξει μέρος από αυτή τη χρηματοδότηση. Και η Πολωνία ήταν ε, ένα παράδειγμα στην κατεύθυνση αυτή, ε, που φελήθηκαν όχι μόνο ο ενεργός πληθυσμός, αλλά και οι φτωχοί από τις αλλαγές. Άρα υπήρχε πρόσβαση, πρόσβαση στην αγορά εργασίας, ε, βελτιώθηκαν ε, το κοινωνικό επίπεδο, ε, η ένταξη στην κοινωνία. Όλα αυτά τα στοιχεία περιλαμβάνονται εις την inclusive growth, η συνολική ανάπτυξη. Ε, δεν θα βοηθήσουμε λοιπόν μόνο εθνικές εταιρείες, αλλά θέλουμε να βοηθήσουμε τους στοχούς. Και σιγά σιγά θα διατυπώσουμε και άλλες προτεραιότητες. Όταν μιλάμε για τη γεωργία, αυτό που είπε ο κύριος Μαρτίνες Μαρτίνες είναι πολύ σωστό και αιτιολογημένο. Έχουμε δηλαδή τομείς τους οποίους εμείς θεωρούμε προτεραιότητες. Την γεωργία, που αναφέρεται στην πράσινη βίβλο και όταν έχουμε προδιαγραφές θα πρέπει οι προδιαγραφές αυτές να εφαρμόζονται και στη γεωργία και στην ενέργεια παραδείγματο χάρη. Μπορούμε ε, να βρούμε ε, διάφορες, ε, διάφορα μικρά βιοποριστικά αγροκτήματα σε άλλους τομείς είναι ίσως τα πράγματα πιο δύσκολα αλλά εφόσον στηρίζουμε τις ανανεώσιμε με πηγές ενεργείας θα πρέπει και οι φτωχοί να υποφεληθούν. Και τέλος, ε, στην ε, έκθεση για την ανάπτυξη σχετικά με το μέλλον της γεωργικής πολιτικής, θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα περιληφθούν αυτά τα στοιχεία στην έκθεση και έχω και εγώ διατυπώσει ορισμένες τροπολογίες. Καλύτερο είναι που συζητάμε εδώ για τη γεωργία στις αναπτυσσόμενες χώρες, αλλά μιλάμε ήδη σε αυτούς οι οποίοι ξέρουν περί τίνος πρόκειται. Εμείς θα πρέπει να φροντίσουμε η δικιά μας γεωργική πολιτική να εφαρμόσει αυτά τα οποία πρεσβεύουμε τόσο στεναρά. Ένα άλλο θέμα είναι η, η αναπτυξιακή πολιτική με, με, ε, εμφανές αποτέλεσμα. Δηλαδή πώς θα μπορέσει να γίνει πιο αποτελεσματική η πολιτική ε, μας. Γνωρίζουμε και τις απαντήσεις, αλλά υπάρχουν και προβλήματα. Θα πρέπει να υπάρχουν ε, μέσα μέτρησης, αξιολόγησης, αλλά δεν θέλουμε να παγιδευτούμε από αυτούς τους δείκτες και από αυτούς, ε, τους, ε, αυτές τις αξιολογήσεις διότι τότε θα επιλέγουμε εύκολες χώρες για να τις βοηθήσουμε όπου θα είναι εύκολο να καταλήξουμε σε αποτέλεσμα να μετρήσουμε τα αποτελέσματα και να τα επιδείξουμε, ενώ άλλες φτωχές χώρες θα παραμείνουν ε, χωρίς βοήθεια. Ε, υπάρχουν λοιπόν ε, μέτρα και σταθμά αλλά δεν πρέπει ε, να περιοριστούμε σε αυτά για να μπορούμε να απευθυνθούμε και σε αυτούς οι οποίοι χρειάζονται πάνω απ' όλα τη βοήθειά μας. Είχαμε και ένα άλλο δίλημα στη συζήτηση. Μυρίσαμε για τις χώρες μετρίου εισοδήματος. Η Επιτροπή μας πήγε στο, στη Βραζιλία, η οποία είναι μια χώρα η οποία θεωρείται σαν ε, χώρα μέσου εισοδήματος και η Ινδία τουλάχιστον στατιστικά. Αλλά οι χώρες αυτές είναι και χώρες όπου υπάρχει ε, ε, όντως ε, βαθιά ένδια. Έχουμε ένα μεγάλο ποσοστό σε αυτές τις χώρες που ζει σε μεγάλη ένδια και θα πρέπει η βοήθειά μας για να αποδώσει να χρησιμοποιείται και σε τέτοιου είδους χώρες. Ε, διότι υπάρχουν και πάρα πολλοί φτωχοί ε, τους οποίους δεν πρέπει να παραβλέψουμε στην περίπτωση αυτή. Για να συνοψίσω τώρα. Η ιδέα στην αρχή ήταν και το αναφέρουμε και σε άλλες εκθέσεις ότι ε, οι επιπρόσθετες, ε, ε, οι επιπρόσθετοι πόροι πρέπει να είναι επιπρόσθετοι και είναι κάτι το οποίο να αντιλαμβανόμεθα πλήρως. Η κυρία Σαργεντίνη σχετικά με την ημερομηνία για τις τροπολογίες. Λέτε ότι η προθεσμία είναι σε δύο μέρες για την έκθεση Κασμάρεκ. 24 ε, Μαρτίου και σήμερα είναι 22. Πολλές φορές η διαδρομή είναι εξίσου σημαντική όπως και η κατάληξη και η γνωμοδότησή σας είναι ο τρόπος ε, με τον οποίο θα επηρεάσουμε την πράσινη ε, βίβλο ε, σχετικά με την αηφόρα ανάπτυξη και την ευρωπαϊκή πολιτική θα έλεγα ότι δεν πρέπει να βιαστούμε να είμαστε πιο επακριβείς κατά τρόπον ώστε να μπορέσουμε να επηρεάσουμε την πράσινη βίβλο διότι εμείς ακόμη δεν έχουμε καταλάβει τι είναι αυτή η inclusive growth, η, ε, ε, αυτό το είδος αναπτύξεως, γιατί να μην επεκτείνουμε λιγάκι την προθεσμία για ε, τις τροπολογίες. Κύριε Ντέβα, συμφωνώ με την κυρία Σαρτζεντίνη. Είναι μια πολύ σημαντική έκθεση και θα έπρεπε να ε, κάνουμε ό,τι χρειάζεται, να καθίσουμε να το σκεφτούμε καλά, να το συζητήσουμε πολύ. Η γραμματεία ε, κάνει την αντίστροφη μέτρηση διότι θα πρέπει ε, να προτείνουμε τις τροπολογίες μας πριν από την αρμόδια επιτροπή, άρα Δευτέρα 28 του μηνός στις 6 το απόγευμα. Δεν βλέπω να υπάρχουν άλλα σχόλια για την έκθεση Κασμάρεκ και δίνω τον λόγο στον κύριο Γκέρχαρτ της Επιτροπής. Pardon, Madam Speaker. Συγγνώμη κυρία Πρόεδρε. Μου δίνετε το λόγο, έτσι. Ναι, έτσι λέει εδώ. Ότι εσείς πρέπει να απαντήσετε. Κάνω λάθος, κάποιος άλλος. Απαντήσαμε τις ερωτηθήσεις ερωτήσεις. Είδε μη, με τα χαρά συνεχίσουμε, να τα καλύψαμε όλα. Δεν ξέρω αν υπάρχουν εκκρεμείς αναπάντητες ερωτήσεις αυτή τη φάση, κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος Τζόνς και η κυρία Σαρτζεντίνη εκ νέου. Συγγνώμη που σας δυσκολεύω τη ζωή. Δεν αναφερόμουν σε χρόνο για άλλη μια έξυπνη τροπολογία, αλλά για μια συζήτηση ακόμα στην Επιτροπή αυτή. Διαφορετικά, αυτή η πράσινη βίβλος μένει αμετάβλητη. Δεν έχουμε περιθώριο αν πάμε στις 28. Δεν έχουμε χρόνο. Νόμιζα ότι τα απάντησε αυτό κύριε Σαρτζεντίνη, λέει η Πρόεδρος. Είπα ότι θα πρέπει να υιοθετήσουμε στην Ολομέλεια ένα ψήφισμα πριν γνωμοδοτήσει η Επιτροπή και μετά θα πρέπει να κάνουμε τις προσαρμογές μέχρι τις 13 Απριλίου. Χρειαζόμαστε 10 μέρες για ε, μετάφραση. Αυτό μπορούμε να κάνουμε. Να απαντήσω σε κάποιες ερωτήσεις που ετέθησαν. Όσον αφορά το χρονισμό, η ανακοίνωση ακολουθεί τις διαβουλεύσεις με θέμα την πράσινη βίβλο. Είχε προγραμματιστεί αρχικά για Ιούνιο. Τώρα μάθαμε ότι ανεβλήθη. Επαόριστον. Δεν έχουμε ημερομηνία. Πιθανότατα αργότερα. Τι να πούμε, Ιούλιο, Αύγουστο. Τώρα, όσον αφορά τις ερωτήσεις. Για αυτή την γενική, τη σφαιρική ανάπτυξη. Υπάρχουν πολλοί ορισμοί όσον αφορά το inclusive growth. Πρότεινε ο κ. Κάσμαρεκ έναν ορισμό. Πώς πρέπει να την αντιληφθούμε, σαν μια ανάπτυξη που καλύπτει όλες τις πληθυσμιακές ομάδες. Όλοι μπορούν να συμμετάσχουν αν εξαιρέσεως και να ωφεληθούν. Έτσι αντιλαμβανόμαστε εμείς αυτή την σφαιρική ανάπτυξη ίσως προταθεί στο μέλλον κάποια πιο ξεκάθαρη, κάποιος ξεκάθαρος ορισμός. Το γιατί προτείναμε αυτή την πράσινη βίβλο την εποχή της διαπραγματεύσεως και τώρα την εποχή αυτή με την οικονομική κρίση τι να σας πω το θέλ, θέλουμε η αναπτυξιακή πολιτική μας να έχει περισσότερα αποτελέσματα έχουμε πέντε χρόνια ή λιγότερα χρόνια στη διάθεσή μας, με νέες σημαντικές προκλήσεις που επηρεάζουν το πρόγραμμα το αναπτυξιακό και αλλάζουν το τοπίο. Αναδύονται νέοι φορείς και μπλεκόμενοι. Κεντρική ιδέα. Η αναπτυξιακή μας βοήθεια πώς θα προσαρμοστεί στην κατάσταση που αλλάζει η συζήτηση όσον αφορά την ενίσχυση, την αποτελεσματικότητά της, πόσο καλά εστιασμένη είναι, αυτά έχω να πω. Θα σταματήσω εδώ. Και αν υπάρξουν άλλες ερωτήσεις, με τα χαράς να απαντήσω. Λοιπόν, λαμβάνοντας υπόψη αυτά τα στοιχεία, η γραμματεία θα επαληθεύσει τις ημερομηνίες και μέσω mail το βράδυ θα σας στείλει την προθεσμία για τις τροπολογίες και η δυνατόν νέα ημερομηνία για τις συζητήσεις. Θα επαληθεύσει ακριβώς τι θα γίνει. Στο σημείο, το σημείο 16. Νέο πρωτόκολλο που καθορίζει τις δυνατότητες αλληλείας και το οικονομικό αντάλλαγμα που βλέπετε από την εταιρική συμφωνία στον αλληλευτικό τομέα μεταξύ Ευρωπαϊκής Ενώσεως και της ε, δημοκρατίας ε, του Σάτομε και Πρίνσιπε. Η κυρία Λεβίν έχει συντάξει ένα σχέδιο γνωμοδοτήσεως. στα πλαίσια του νέου πρωτοκόλου αλλιές μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και της μικρής δημοκρατίας ε, Έχετε το λόγο κυρία Λεβίν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα, η συμφωνία, η προηγούμενη συμφωνία έληξε στις 31 Μαΐου 2010. Το νέο πρωτόκολλο εφαρμόζεται προσωρινά Μέχρι να ε, ολοκληρωθεί η διαδικασία έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το νέο πρωτόκολλο θα ισχύει για τρία χρόνια. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε μπορεί να εγκρίνει είτε να απορρίψει αυτό το πρωτόκολλο. Θα ήθελα να αναφέρω την αλλιευτική συμφωνία με την Μαυριτανία που θα συζητηθεί στην Ολομέλεια την επόμενη σύνοδο. Όπως ξέρετε, η αλληλευτική πολιτική, η πολιτική είναι θέμα συναπόφαση. Όσον αφορά τα αλληλευτικά πρωτόκολλα, οι συμφωνίες, εμείς μπορούμε μόνο να συνενέσουμε, δεν μπορούμε να αλλάξουμε τίποτα και δεν μπορούμε να τροποποιήσουμε τις συμφωνίες αυτές. Στην Επιτροπή Ελίας αναλάβαν την πρωτοβουλία να προσπαθήσουμε να ε, συμμετέχουμε σε μία πρώτη φάση των διαπραγματεύσεων κάνοντας τις ε, ε συμμετέχοντας κάνοντας τις μας Ανέφερα την Μαυριτανία δεδομένου ότι πρόκειται για την έκθεση που θα ψηφιστεί στην επόμενη Ολομέλεια στο Στρασβούργο. Τι θέλουμε να κάνουμε τώρα, να εξασφαλίσουμε ότι οι συμφωνίες αυτές ευθύς εξ αρχής αναφέρουν τις αρχές οι οποίες θέλουμε να ακολουθηθούν και θέλουμε οι μηχανισμοί να εφαρμοστούν όπως πρέπει. Οι μηχανισμοί που προβλέπονται. Τώρα, όσον αφορά αυτή την ε, αλληλευτική συμφωνία με τη μικρή αυτή χώρα, το Σάουτο με Πρίνσιπε. Μιλούμε για 2.047.500 εκατομμύρια ευρώ κοινοτική χρηματοδότηση για 7.000 τόνους που αντιστοιχεί σε 40 λιευτικά σκάφη που αλλιεύουν στα είδατα του Σότομε και πριν είπε τόνο. Θεσπίζεται στη συμφωνία ότι μπορούν λοιπόν να αλλιευθούν 7.000 τόνοι τουλάχιστον, δεν υπάρχει ανώτατο όριο, Εάν λοιπόν ο αλλιευτικός στόλος είναι τυχερός, μπορούν να αλλιεύσουν βάσει της συμφωνίας και ε, μεγαλύτερες ποσότητες, καταβάλλοντας κάποιο τίμημα βεβαίως. Κάτι άλλο το οποίο νομίζω ότι πρέπει να ενδιαφέρει το Κοινοβούλιο είναι το θέμα της πρόσβασης του Κοινοβουλίου στην αξιολόγηση αυτής της συμφωνίας. Διότι, εάν συνενέσουμε για τη συμφωνία αυτή, Νομίζω ότι είναι λογικό να ζητήσουμε πριν να συνενέσουμε να έχουμε πρόσβαση στην όλη αξιολόγηση, να δούμε πώς λειτουργήσαν και στο παρελθόν παρεφέρει συμφωνίες. Μέχρι πριν από δύο μήνες αποφάσισε η Επιτροπή να μας δώσει περιορισμένη πρόσβαση, διότι έχουν διαβαθμίσει τις πληροφορίες. Εμείς, εγώ λοιπόν για να έχω πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα θα πρέπει να πάω στη γραμματεία, να περιμένω, υπογράψω ένα χαρτάκι, να κάνω αίτηση και μετά να μην μπορώ να παίρνω σημειώσεις, απλώς να διαβάσω. Εάν λοιπόν πρόκειται για εμπιστευτικές προφορίες, θα πρέπει εγώ να προσπαθήσω να θυμηθώ κάποια πράγματα, αλλά κάποια δεν μπορώ παρά να τα περιλάβω εδώ. Έχετε λοιπόν ε, περιορισμένοι ε, πιστευτικές πληροφορίες στη σελίδα 4 και στη σελίδα 3, οι οποίες ε, είναι στις παραγράφους που έχουν το bullet point στην αρχή. Έχουμε να κάνουμε τώρα με μια πάρα πολύ μικρή και φτωχή χώρα που έχει το μεγαλύτερο εισόδημά της από την Αλία για λόγους υγειονομικούς δεν μπορεί να εξάγει τα αλλιεύματά της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, στην Αμερική, με συγχωρείτε. Σύμφωνα με... Ίσως ξέρετε ότι ένα μέρος του ποσού που δίδεται σε τέτοιου είδους συμφωνίες δίδεται για να ενισχυθεί ο έλεγχος ε, της αλίας, ε, να ληφθούν τα κατάλληλα διοικητικά μέτρα, να γίνουν οι σωστές έρευνες, η σωστή επιθεώρηση, που είναι πάρα πολύ περίεργες εμβέλειες σε εθνικό επίπεδο στη χώρα αυτή. Κάτι άλλο που βρήκε στις πληροφορίες είναι και εν πάση περιπτώσει κατά κάποιο τρόπο είναι καλές αυτές οι συμφωνίες. Γιατί αν η Ευρωπαϊκή Ένωση μια είδους, έχει μια τέτοιου είδους ε, εκκρεμή συμφωνία με τις χώρες αυτές σημαίνει ότι ο ιδιωτικός, κανένας ως ιδιώτης δεν μπορεί να ε, συνάψει συμφωνίες μόνο ό,τι μπορεί να κάνει μπορεί να το κάνει στα πλαίσια αυτών των κοινοτικών συμφωνιών. Επίσης πρέπει να πω ότι υπάρχουν και κάποιοι Ευρωπαίοι οι οποίοι αλλιεύουν στα ύδατα του Σάτομε Πρίνσιπε με άλλη σημαία, πράγμα το οποίο δεν ε, πρέπει να γίνει ε, αποδεκτό, δεδομένου ότι έχουμε αποκλειστικέ συμφωνίε τέτοιου είδου καταστάσεις δεν πρέπει να συμβαίνουν. Επίση, στην ε, συμφωνία αυτή λέγεται ότι θα πρέπει να υπάρχουν κατάλληλε εγκαταστάσεις για την φόρτωση εκφόρτωση για τις εκφορτώσεις να γίνεται προσπάθεια να ε, υπάρχουν νέες θέσεις απασχόλησης στον τομέα. Όσον αφορά τα αποθέματα και το περιβαλλοντικό θέμα, κάποιες από τα αποθέματα, κάποια είδη τόνου, Ε, και άλλα αλλιευόμενα ήδη μας απασχολούν, καθώς και το υπάρχουν ανησυχίες για τα παρεπίπτοντα αλλιεύματα. Επίσης υπάρχουν χώρες Λέγουν με αυτού του είδους τις συμφωνίες δίδει και μεγάλη υποστήριξη στις εθνικές αρχές. Η συνεισφορά στις αρχές, σύμφωνα με την, που ασχολούνται με τον αλληλευτικό τομέα, και η στήριξη αφορά την κατάρτιση νεολογίου, τα συστήματα ελέγχου για τα σκάφη που αλλιεύουν και παρά το γεγονός ότι δεν έχει υπάρξει πολύ μεγάλη πρόοδος, υπάρχει μια κάποια πρόοδος και κάποιες επιτεύσεις με την κοινοτική χρηματοδότηση. Δύο πράγματα θα ήθελα να προσθέσω για την αξιολόγηση αυτή. Πρώτα απ' όλα, ότι δεν θα πρέπει τέτοιες πληροφορίες να είναι διαβαθμισμένε δεδομένου ότι καθίσταται πάρα πολύ δύσκολο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να κάνει σωστά τη δουλειά του, εάν δεν έχει πρόσβαση σε αυτά τα έγγραφα. Είχαμε στο παρελθόν ε, πρόσβαση σε αυτά τα έγγραφα. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει το θέμα αυτό να το συζητήσουμε και να αντιταχθούμε σε τέτοιου είδου πρακτικέ, πράγμα που έχει γίνει στο παρελθόν στην Επιτροπή Ελία. Τώρα, όσον αφορά την ε, αξιολόγηση, νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχουν πολύ σαφή κριτήρια όσον αφορά τη γνωμοδότηση. Δηλαδή, εάν όντως ε, οι συμφωνίες αυτές είναι συμφωνίες που λειτουργούν όπως θα έπρεπε. Όσον αφορά τις συστάσεις. Πολλά θα πρέπει να γίνουν όσον αφορά την διαφάνεια για το σύνολο επίσης των αλλιευμάτων διότι δεν γνωρίζουμε ποιε είναι οι ανώτερε ποσότητες αλλιευμάτων. Νομίζω ότι όλα αυτά θα πρέπει να αποτελούν αποτέλεσμα διαφωνών διαδικασιών. Ξέρω ότι υπάρχουν συναντήσεις μεταξύ της ε, Κομισιόν και των χωρών και πιστεύω ότι τέτοιου είδους συμφωνίες θα πρέπει να παρακολουθούν εκ των για να δούμε πώς χρησιμοποιούνται τα κοινοτικά κονδύλια όταν υπάρχουν τέτοιου είδους συμφωνίες. Επίσης, τα θέματα διαχείρισης των ε, αλλιευμάτων και το θέμα της ύπαρξης ε, ε, κάποιων παρατηρητών για ενημέρωση δεν έχουν γίνει ε, συμβατά. Επίσης, όσον αφορά την ε, αρχή της αποκλειστικότητας, θα πρέπει αυτή να τηρείται. Η εφαρμογή αυτής της συμφωνίας ε, επίσης θα πρέπει να αποτελεί αντικείμενο της ίων αναφορών που θα υποβάλλονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με διαφάνεια. Αυτές ήταν οι κυρίες παρατηρήσεις που θέλω να κάνω. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ντέβα έχει το λόγο. Thank you, Madam Chairman. Mrs. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Έξοχα αυτά που μας είπε η κυρία Λοβέν. Και συνεχώς κάνουμε αυτό που κάνουμε. question, Madam Chairman. Ερώτηση, κυρία Πρόεδρε. Στο λαό τους ε, Σαν Τομέ και Πρίνσιπε, τους δίνουμε 2 εκατομμύρια ευρώ για να προστατεύσουν 7.000 τόνους τόνου. Αν τηρήσουμε κατά γράμμα τη συμφωνία, ούτε ένας τόνος παραπάνω από τις 7.000 τόνους δεν αφαιρείται, τηρούμε τη συμφωνία στο γράμμα του νόμου. Γιατί υπογράψαμε. Ερώτηση τώρα. Ποια είναι η αξία των 7.000 τόνων τόνου του ψαριού στην αγορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 245, 245 εκατομμύρια ευρώ, παρακαλώ. So we give them million. Τους δίνουμε 2 εκατομμύρια ευρώ και τα πουλάμε για 245 εκατομμύρια ευρώ. That's why keeping the figures secret. Γι' αυτό παραμένουν μυστικά τα νούμερα. Έτσι. Είναι δίκαιο, είναι σωστό. Είναι εκμετάλλευση ή δεν είναι. Τι είναι αυτό, πώς θα το πούμε. Πώς το δικαιολογούμε. Αρσένης. Ποιος Αρσένης. Merci Συμφωνώ με τον κύριο Ντέβα. Για τα στοιχεία ίσως είναι ακόμα πιο υψηλά τα ποσά. Η αξία του, του τόνου στην αγορά στην Ευρώπη. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένα από τα προβλήματα η εκμετάλλευση. Είναι ένα από τα προβλήματα αυτών των συμφωνιών. Άλλο πρόβλημα. Αυτά που μας είπε η κυρία Λόγαν ήταν, ήταν πολύ σωστά, ήταν πληρέστατα τα σχόλιά της. Είναι σημαντικό ότι αυτοί οι άνθρωποι χρειάζονται το ψάρι για να το φάνε. Τους παίρνουμε το ψάρι, τα ψάρια τους και οι μικροί ψαράδες βλέπουν τα μεγάλες τις μεγάλες βάρκες, τα μεγάλα πλοία να τους παίρνουν τα ψάρια τους. δεν βελτιώθηκε η βιώσιμη αλία, δηλαδή η βιώσιμη διατροφή τους από την αλία. Δεν παίρνουμε το πλεόνασμα του αλλιευτικού αποθέματος. Δεν έχουμε κάνει αποτίμηση του αλλιευτικού αποθέματος να δούμε πόσα ψάρια, τι ψάρι χρειάζονται οι ντόπιοι, τι βάρος και να δούμε τι απομένει και αλλιεύουμε με βιώσιμο τρόπο εμείς. Και συνεχίζεται αυτή η κατάσταση. Δεν υπάρχουν έλεγχοι. Οι υπεύθυνε επιτροπές που πρέπει να υποπτεύουν σωστή εφαρμογή των συμφωνιών δεν συνεδριάζουν. Και τα προβλήματα αυτά είναι κοινά προβλήματα σε όλες αυτές τις αληθικές συμφωνίες. Και εδώ προστίθεται και άλλο θέμα. η ταξινόμηση των αξιολογήσεων. Κάτι που δημιουργεί νέες δυσκολίες στο έργο του Κοινοβουλίου. Και πρέπει να δώσουμε σύμφωνη γνώμη μετά από την θέση σε ισχύ αυτών των συμφωνιών. Και αυτό είναι άλλο ένα πρόβλημα που προστίθεται. Χάλια κατάσταση. Ποια είναι η αλήθεια. Αν δεν συνάψουν συμφωνίες με αυτές τις χώρες, άλλες χώρες με πολύ λιγότερο βιώσιμες πολιτικές θα συνάψουν συμφωνίες. Εγώ δεν είμαι κατά των αληφτικών συμφωνιών, αλλά πρέπει να αλλάξει ριζικά το περιεχόμενο των συμφωνιών μας. Σημαντικό στοιχείο όλων αυτό. Κάτι που ενδιαφέρει πολύ την Επιτροπή μας. Η αναπτυξιακή πτυχή των συμφωνιών αυτών πάντα υπονομεύεται. Και η έκθεσή μας θα πρέπει να εστιάζεται πολύ σε αυτό. Διότι είναι πολύ σημαντικό θέμα. Η έλλειψη βιωσιμότητας όσον αφορά την προσέγγιση που ακολουθούμε για την σύναψη αυτών των συμφωνιών. Οι δεσμεύσει που έχουμε αναλάβει όσον αφορά την ανάπτυξη. ονομαστικά πληρούνται και μόνο. Και αν πληρούνται. Ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω το λόγο στον εαυτό μου, λέει Πρόεδρος. Ξέρω το Σάουτο Μέ και Πρίνσιπε, διότι βοήθησα την κυβέρνηση να καταπολεμήσει τη διαφθορά, να διευρύνει τις οικονομικές αποκλειστικές δραστηριότητες της είναι μια χώρα που δεν έχει σχεδόν καθόλου δρόμους, δεν έχει πανεπιστήμιο, ένα λύκειο έχει. Δεν έχει ακτοφυλακή. Όλα τα δικαστικά συστήματα, το δικαστικό σύστημα αποτελείται από 16 άτομα. Είναι πάρα πολύ στερημένη. Και δεν βλέπω πώς θα μπορούσαμε με κάποιο τρόπο να διαπιστώσουμε ότι αυτές οι συμφωνίες θα γίνουν σεβαστές. Ίσως θα μπορούσαμε να καλέσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας πει ποια μέτρα αναπτυξιακής βοήθειας ε, θα μπορούσαν να τους βοηθήσουν να δημιουργήσουν συστήματα ελέγχου. Αυτές οι συμβάσεις δημιουργούν τεράστια προβλήματα, πράγματι, και αυτό πάντα με ενοχλεί. Έχουν τη σφραγίδα της ανάπτυξης αλλά το αντίθετο επιτυγχάνουν. Το ακριβώς αντίθετο. Αυτά ήθελα να σας πω. Είναι μια χώρα που έχει μία πτήση την εβδομάδα που ξεκινά, φεύγει από Λισαβόνα. Πολύ απομονωμένη χώρα, πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Και δεν είναι σε θέση να ελέγξουν το παραμικρό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει το λόγο. Ο κ. Αλεξάνδρου έχει το λόγο. Merci, Madame la Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Συμφωνώ απολύτως με την περιγραφή σας της κατάστασης ε, του Σαοτόμ ε, και Πρεντσιπέ και δεν έχω τίποτα να προσθέσω. Όσον αφορά την παρουσίαση την οποία έκανε η κυρία Λεβίν, προσωπικά τη βρίσκω πολύ ενδιαφέρουσα γιατί μας επέτρεψε να δούμε ορισμένες ε, πτυχές ε, τις οποίες το νέο πρωτόκολλο θα έπρεπε να οδηγήσει σε μία βελτίωση της κατάστασης. Εάν λοιπόν μου δώσετε τη δυνατότητα να αναπτύξω περισσότερο τα θέματα αυτά και μετά θα επανέλθω σε σχόλια των άλλων ε, ε, Ευρωβουλευτών μιλάμε για μια συμφωνία για τον τόνο και το πρωτόκολλο αναφέρεται εις τα αλλιευτικά τα οποία μπορούν ε, να καλύπτουν μια τονοχωρητικότητα αναφοράς αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις δεν επιτυγχάνεται, δεν γίνεται σεβαστό το πρωτόκολλο αυτό. Λοιπόν, έχουμε ήδη μία ε, πληρωμή για να έχουμε πρόσβαση εις ε, την, στο ε, προϊόν γιατί υπάρχει μεταφόρτωση του προϊόντος και για να μπορέσουμε να να ψαρεύουν ε, ε, τα πλοία αυτά ε, χρειάζονται μεγάλο χώρο και γι' αυτό προσπαθούμε να συνάψουμε συμφωνίες αλληλείας με τις παράκτιες χώρες. Αυτό είναι το ένα θέμα. Επίσης πρέπει εμείς σαν Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν προσπαθούμε να διαπραγματευτούμε με μια τρίτη χώρα η οποία δεν έχει την κατάλληλη υποδομή για να μπορέσει να παρακολουθήσουμε τις δραστηριότητες των πλοίων μας, να εξασφαλίσουμε ότι η στήριξη του τομέα και το ποσοστό της χρηματοδότησης που απευθύνεται στην αλληλεία θα μπορέσει όντως να φτάσει στον τομέα της αλληλείας διότι παραδείγματο χάρη όλοι αναφέρατε και είπατε ότι οι αρχές του ΣΑΟ δεν είναι σε θέση να ελέγξουν τις δραστηριότητες. Συμφωνούμε, το είπατε κι εσείς. Δεν υπάρχει η υποδομή, δεν υπάρχουν ακτοφύλακες και μέσω αυτού του πρωτοκόλλου το οποίο έχει εκπνεύσει προσπαθήσαμε να καταρτήσουμε στο ΣΑΟ το σύστημα VMS το οποίο είναι τεράστιο σε σχέση με την κατάσταση στην οποία βρισκόταν η χώρα. Βεβαίως θα μου πείτε ότι το VMS δεν είναι το σύμπαν, αλλά θα επιτρέψει το σύστημα αυτό να παρακολουθούμε τις δραστηριότητες των πλοίων, των αλευτικών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως αλλά και των άλλων πλοίων ε, εφόσον ε, έχουν ε, αυτόν τον μηχανισμό ανιχνεύσεως και πάνω σε μία οθόνη θα παρακολουθεί κανείς την ε, ε, κίνηση των πλοίων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, πράγμα το οποίο θα επιτρέψει να ε, συνδυάσει κανείς και από εκεί να καταλάβει ποιες είναι οι ποσότητες των αλλιευμάτων. Και έτσι οι τοπικές αρχές θα μπορέσουν να επέμβουν και να παρακολουθούν αυτά τα πλοία. Ε, με το νέο πρωτόκολλο λοιπόν θα προσπαθήσουμε να συνεχίσουμε να χρηματοδοτούμε αυτές τις απαραίτητες μεθόδους για την παρακολούθηση της αλληλείας. Επίσης μιλήσατε για τους παρατηρητές. Σας ε, υπενθυμίζω ότι το κείμενο του πρωτοκόλλου και το παράρτημα προβλέπει ότι οι παρατηρητές μπορούν να ε, επιβαίνουν στα πλοία κατόπιν ετήσεως των αρχών του ΣΑΟΤΟΜΕ, πράγμα το οποίο δεν πράττουν οι αρχές. Και γιατί δεν το πράττουν, διότι δεν υπάρχουν παρατηρητές. Θα έπρεπε λοιπόν κάποιο σχόλιο. Ο κύριος Αλεξάνδρου λέει θα προτιμούσα να μην απαντήσω σε αυτή την ερώτηση. Θα έπρεπε λοιπόν στο επόμενο πρωτόκολλο όσον αφορά τη στήριξη του κλάδου να προβλέψουμε μέτρα σύμφωνα με τα οποία οι παρατηρητές θα εκπαιδευτούν και κατά συνέπεια στη συνέχεια θα μπορούσαν να ε, ε, επιβαίνουν των πλοίων. Επίσης, θέλω να σας υπενθυμίσω ότι τα αλλιευτικά τόνου δεν αλλιεύουν εκεί όπου αλλιεύουν και οι ε, χειρονακτικοί, τα χειρονακτικά ε, και απλά αλλιευτικά, αλλά μετά τα 12 μίλια και το VMS θα μπορέσει να επαληθεύει ανα πάσα στιγμή αν αυτό ευσταθεί ή όχι. Αυτό λοιπόν στο οποίο αποβλέπουμε για τα βαπόρια της Ευρωπαϊκής Ενώσεως είναι ε, ε, ε, είναι αλλιευτικά τόνου που δεν έχουν ε, καμία σχέση με την αλλίευση των ε, απλών ψαριών που προσφέρουν πρωτεΐνες ή στον πληθυσμό των παρακτήων χωρών. Επίσης ζητήσαμε από τις αρχές του ΣΑΟΤΟΜΕ να προτείνουν πληρώματα αυτόχθονα που θα μπορούσαν να επιβιβαστούν των αλλιευτικών. Αυτοί όμως προτιμούν ε, να έχουν πληρώματα από χώρες ΑΚΕ με ένα ποσοστό υπηκών του ΣΑΟΤΟΜΕ. Και αυτά είχα να σας πω. Βέβαια είναι προφανές ότι το πρωτόκολλο όπως έχω, τα έχουμε διαπραγματευτεί στο παρελθόν θα πρέπει να βελτιωθούν. Ελπίζουμε δε ότι το πρωτόκολλο αυτό ακόμη και εάν δεν μπορεί να θεωρηθεί πανάκια θα ακολουθεί την, ε, ε, την μέθοδο που διέπει τις σχέσεις μας με τις ε, χώρες αυτές για να αναπτυχθεί η αλληλεία τους και να υπάρχει μια συγκεκριμένη αξία και μια ποιοτική βελτίωση. Αντιλαμβάνουμε τις ανησυχίες των ΜΕΝ και των ΔΕ σχετικά με την την ιολόγηση αλλά αντιλαμβάνεστε ότι είναι κάτι το οποίο εγώ δεν μπορώ να παρακολουθήσω γι' αυτό και θα προσπαθήσω να, να ε, ε, μεταβιβάσω εις ε, τις υπηρεσίες μου τα, τις ανησυχίες σας μέχρι τώρα. Η κυρία Λέβιν έχει το λόγο για να ολοκληρώσει. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για τα σχόλια και τις παρατηρήσεις που συμμερίζουμε και να ευχαριστήσω τον κύριο Αλεξάνδρου εκ μέρους της Επιτροπής. Διότι είπε καλόπιστα ότι θα πρέπει να έχουμε καλύτερη συμφωνία στο μέλλον. Ίσως εγώ δεν ήμουν απόλυτα σαφής για τον τρόπο με τον οποίο θα εξασφαλίσει ε, καλύτερη υποστήριξη στον τομέα αυτό, καλύτερες συμφωνίες στο μέλλον η Κομισιό. Το θέμα της διαφάνειας των ετησίων εκθέσεων, κοινών συναντήσεων με την Επιτροπή είναι θέματα τα οποία επίσης θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και να είμαστε σίγουροι ότι υλοποιούνται όλες αυτές οι καλές προθέσεις που έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το θέμα των παρατηρητών μου προκαλεί μια κάποια σύγχυση. Εγώ δεν πρέπει να διαβάσω την αξιολόγηση, διότι λέγεται ότι μέχρι τώρα δεν έχουν υπάρξει ε, παρατηρητές, πράγμα το οποίο δυσαρεστεί και τις αρχές του Σάου Τομέ Πρίνσιπε, παρά το γεγονό ότι είναι δύσκολο εκ των προτέρων να γίνει μια τέτοια πρόταση. Σήμερα λοιπόν με την αξιολόγηση λέγεται ότι οι διάφοροι οικονομικοί κοινοτικοί φορείς δεν μπορούν να δώσουν την κατάλληλη ενημέρωση τους παρατηρητές αρκετά έγκαιρα, άρα υπάρχει δυσαρέσκεια που εκφράζεται το θέμα αυτό εκ μέρους των ορχών του ΣΑΟΤΟΜΕ. Τώρα σαν αφορά την περίπτωση του κ. Ντέβα για την αξία, την εμπορική αξία των αλλιευμάτων. Είπαμε ότι πρόκειται για μία χώρα η οποία έχει ένα φυσικό αλλιευτικό πόρο, πάρα πολύ φτωχή, που δεν μπορεί να κάνει μόνη της την εξαγωγή αυτού του λευτικού πόρου που διαθέτει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βεβαίω χρειάζεται να, γίνεται και, να υπάρξει και υποστήριξη και επιτήρηση, αλλά θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί ώστε να γίνονται σωστά τα πράγματα. Αυτό είναι κάτι το οποίο λέγεται και στην αξιολόγηση. Δεδομένου ότι πρόκειται, η Αλία είναι μία πάρα πολύ σημαντική πηγή ε, απασχόλησης. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι υπάρχει ίσως κάποια σημαντική παρανόηση. Μας είπατε ότι το ΣΑΟΤΟΜΕ δεν έχει παρατηρητές και στην έκθεση αναφέρεται ότι δεν μπορούν να επιβιβάζονται στα πλοία οι παρατηρητές. Υπάρχει αντίφαση εδώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Νομίζω ότι στην παρέμβασή μου ξέχασα να τονίσω το θέμα της διαφάνειας. Όντως, θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι στο παρελθόν υπήρχε πρόβλημα με την διαφάνεια. Αυτό το οποίο προβλέπεται και η κυρία Λέβιν επέκρινε τις υπηρεσίες της Κομισιόν στον Ειρηνικό, που δεν τήρησαν τις ε, υποχρεώσεις της ε, μικτής επιτροπής, όχι μόνο εγώ, αλλά και όλοι στην υπηρεσία μου συμφωνήσαμε ότι θα πρέπει να τηρούνται οι κανόνες διαφάνειας. Θα γίνει αυτό και είχα πει πέρσι στο τέλος του χρόνου ότι αυτό είναι κάτι το οποίο θα γίνει συστηματικά. Δηλαδή, υπάρχει μια ετήσια μεικτή συνάντηση της Μεικτής Επιτροπής που κάνει την αξιολόγηση της αξιολ... την, ε, συγγνώμη, την αξιολόγηση τέτοιου είδους ε, ε, συμφωνιών. Χωρίς λοιπόν να υπάρχουν οι εργασίες αυτής της Μεικτής Επιτροπής, δεν μπορεί να γίνει τίποτα και συμφωνώ απόλυτα με αυτά που είπε η κυρία Λέβιν. Όσον αφορά τώρα τους παρατηρητές, υπενθυμίζω ότι το κείμενο του παραρτήματος διευκρινίζει ότι αυτό γίνεται αιτήση των αρχών του ΣΑΟΤΟΜΕ. Τώρα, πώς, τι σημαίνει αυτό στην πραγματικότητα, υπάρχουν οι σχετικές ε, διατάξεις. Εάν το ΣΑΟΤΟΜΕ παρατηρήσει ότι τα πλοία αρνούνται να επιβάσουν ένα παρατηρητή, είναι πολύ σαφή τα πράγματα. Για την επόμενη ελευτική περίοδο δεν θα πρέπει να χορηγείται στα σκάφη αυτά άδεια για να υποστεί κύρωση στο σκάφος το οποίο δεν θέλει να επιβιβάσει τον παρατηρητή. Τους δίδεται αυτή η δυνατότητα. Επίσης είναι πολύ ενδιαφέρουσα η παρατήρηση της κυρία Λέβιν για τις προτεραιότητες που πρέπει να καθοριστούν στα πλαίσια της υποστήριξης του κλάδου και κυρίως να βελτιωθούν οι φυτογειονομικές καταστάσεις ότι οι εξαγωγές αλληλευτικών προϊόντων από το ΣΑΟ πριν πρίνσιπε να μπορέσουν να φτάσουν στη κοινοτική επικράτεια. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να συζητηθεί μεταξύ, τους, μεταξύ μας. Και θα είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το διαπραγματευτούμε μεταξύ τους, διότι όλα αυτά πρέπει να γίνουν στα πλαίσια της επόμενης Μικτής Επιτροπής, ώστε τα κονδύλια που προβλέπονται για αυτό το συγκεκριμένο στόχο να συνεισφέρουν πραγματικά στην ενίσχυση του μέλλα. Συμφωνώ απόλυτα με την παρατήρηση της κυρίας Λέβη. Ευχαριστώ. Λοιπόν, προθεσμία κατάθεση τροπολογιών 30 Μαρτίου 12 η ώρα το μεσημέρι. Ψηφοφορία θα λάβει η χώρα στις 2 Μαΐου. Περνάμε στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διαταξής που αφορά τη χρηματοδότηση ενίσχυση υποδομών φραγμάτων σε αναπτυσσόμενες χώρες. Έχει συντάξει ένα σχέδιο έκθεσης ο κύριος Ντέβα για την διαχείριση των ειδεπίτων πόρων, την επιβίωση των πληθυσμών που ζουν στα Ιμαλάγια μεταξύ άλλων και τις αβεβαιότητες που... Λοιπόν, για αυτούς που δίνουν χρήματα είναι το θέμα οικοδόμηση φραγμάτων όσον αφορά του παγετώνε και είναι πολύ σημαντικό για κοινωνικέ συνέπειε, περιβαλλοντικέ συνέπειε, για κάποιε αναπτυξιακέ δράσει στον τομέα των υποδομών. Λοιπόν, κύριε Ντέβα, έχετε το λόγο ούτω ώστε να παρουσιάσετε την έκθεσή σα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για αυτή την εισαγωγή αυτή η έκθεση πέρασε μεγάλη περίοδο διότι αφορούσε περιβάλλον και ανάπτυξη αρχικά και κατέληξε με ενίσχυση των διαφόρων υποδομών φραγμάτων. η Επιτροπή Περιβάλλοντος θεώρησε ότι ήταν εντολή της να μιλάει για το περιβάλλον και δεν είχε σχέση με την Επιτροπή Ανάπτυξης. Έπρεπε λοιπόν να είμαι προσεκτικό όσον αφορά τον τίτλο της εκθέσεως. Όμως το θέμα είναι απλούστατο. Οι παγετώνες στις μεγάλες ορεινές περιοχές συμπεριλαμβανομένων των Ιμαλαίων λιώνουν γρήγορα. Όχι λόγω αύξησης θερμοκρασίας, θα μπορούσε να είναι και αυτό το αίτιο και αυτό συμβάλλει, αλλά η βασική, ο βασικός λόγος, αναμφισβήτητος λόγος, αίτιο, που λιώνουν πιο γρήγορα οι παγετώνες από το αναμενόμενο είναι λόγω εθαλομίχλης από, τις, ε, από τα μαγείρια, από τις κουζίνες που χρησιμοποιούν ε, κάρβουνο, από το μαύρο άνθρακα. Πολλές χώρες της Άνδης και γύρω στα Ιμαλάια ε, και είναι ξύλα στους φούρνους τους για να ψήσουν το φαγητό. Και ο καπνός ανεβαίνει στην ατμόσφαιρα και θαλομίχλη, μικρά κομμάτια άνθρακο, μόρια, πάνε και να αποτίθενται στο χιόνι. Άμα πέσει το φως του ηλίου, στο μαύρο, καταλαβαίνετε τι γίνεται. Περνάει η ακτίνα και αρχίζει να λιώνει το, τον πάγο. Εξ αυτού λοιπόν, είχαμε επιτάχυνση της τήξης των πάγων και συλλογής ύδατος. Όχι γύρω από τα φράγματα που είχαν κατασκευαστεί, που ήταν ανθρώπινες κατασκευές, αλλά γύρω από φράγματα που έφτιαξε η φύση. Χωρίς ενίσχυση στις, πλευρές, στις όχθες, στις ούτε στα, στις πλευρές των φραγμάτων. Μιλάμε για μεγάλα κενά ε, συρροής, ε, μεγάλα, μεγάλες βλάκους συρροής υδάτων φυσικούς. Έγινε πολύ μεγάλη έρευνα από την Μότ και άλλους και στο Νεπάλ και αλλού και είπαν ότι περίπου 200 φράγματα πάνω κάτω υπάρχουν σε αυτή την περιοχή, τώρα που κουβεντιάζουμε, που θα μπορούσαν να σπάσουν. Διότι είναι φυσικά φράγματα. Στο, στο κόλμο Ρέγκς δεν πήγε κάποιος και το έφτιαξε. Έχει συλλεγεί πολύ νερό εδώ και όπως ισορεύεται και κατεβαίνει το νερό, δημιουργεί αστραπίες πλημμύρες, τεράστια καταστροφική δύναμη από το νερό παρασύρει χωριά, το νερό και ό,τι θέλετε. Και αυτό επιταχύνεται. Κανείς δεν το πρόσεξε πόσο συχνά συμβαίνει μέχρι πρόσφατα ε, στο Πακιστάν. Στο Νεπάλ, στο Πακιστάν. Και, και τα Ιμαλάια είναι σε περιοχή σεισμογενή. Και αν γίνει σεισμός όπως αυτός που συνέβη στην Ιαπωνία, σε αυτή την περιοχή, καταστροφή θα είναι κάτι φάνταστο, το αδιανόητο. Όχι μόνο θα εξαφανιστούν οι υδάτινοι πόροι, θα εξαφανιστούν και χωριά. Το είδαμε στο Πακιστάν. Θα μπορούσε να εμποδιστεί, να προβλεφθεί και δεν έγινε τίποτα. Δεν είναι μόνο θέμα τυχαίο αυτό. Αν συμβεί αυτό, τα ποταμοί που τροφοδοτούν αυτή την περιοχή τροφοδοτούν 1,5 δισεκατομμύριο ανθρώπους στα μεγάλα ποτάμια, μέσα των μεγάλων ποταμιών της Ασίας. Θα αλλάξουν νερού, αν συμβεί αυτό, και αυτό έχει τεράστιες συνέπειες όσον αφορά τη γεωργία της περιοχής του κόσμου αυτής. Μιλάω για δισεκατομμύρια ανθρώπων που θα πεινάσουν. Άρα έχουμε συνδυασμό παραγόντων Σεισμός, δυνατότητα σεισμού. Να σπάσουν τα φράγματα. Λιώνουν πιο γρήγορα το προβλεπόμενο οι παγετώνες. Και ο άνθρακας, τα σωματίδια του άνθρακα που εξακολουθούν να πέφτουν, κάνει κανείς τίποτα απ' όλα για όλα αυτά. Και το χειρότερο, είναι μια περιοχή που αποτελείται από τον Μπουτάν, τον Νεπάλ, το Πακιστάν, την Ινδία και την Κίνα. Επισκέφθηκα την περιοχή με ελικόπτερο στα 18.000 πόδια για να δω όλα αυτά τα οποία σας παρουσιάζω σήμερα. Κανείς δεν έχει καθίσει γύρω από ένα τραπέζι να κουβεντιάσει το θέμα του νερού, το θέμα των φραγμάτων, διότι οι Πακιστανοί και οι Ινδοί και οι Κινέζοι δεν μπορούν να μαζευτούν να κουβεντιάσουν ούτως ή άλλως. Δεν κάθονται μαζί. Στην έκθεση ζητώ μια διεθνή υπηρεσία, ίσω υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, να δημιουργηθεί και να μπορέσουν να καθίσουν να συζητήσουν αυτό το θέμα. Δεν είναι κάτι που η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να φιλοξενήσει, διότι θα αναρωτιόταν οι πάντε τι δουλειά έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ. Θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε όμω τον ΟΗΕ να δημιουργήσει αυτό το φορέα. Και έχουμε αυτή την έξοχη ερευνητική οργάνωση που ξεκίνησε από πολύ καλού Νορβηγού, Σουηδού και Ευρωπαίου επιστήμονε σε αυτή την περιοχή του κόσμου που εξεπώνησαν διαδοχικά πολλές εκθέσεις. Κανείς δεν έδωσε τη δέουσα προσοχή. Λόγω της περιφερειακής πολιτικής, πολιτικών παιχνιδιών μεταξύ Πακιστάν, Ινδίας και Κίνας. Αντιμετωπίζουμε μια απειλή. Εκατό φορές χειρότερη απειλή από αυτή που είδαμε στην Ιαπωνία. Και θέλω να ξεκινήσουμε μια συζήτηση Δηλαδή, πώς να το αποφύγουμε αυτό. Να αποφύγουμε να συμβεί αυτό. Διαφορετικά εκατομμύρια εκατομμυρίων άνθρωποι θα πεθάνουν και θα πεθάνουν και από την πείνα. Ευχαριστώ πολύ λοιπόν. Είμαι ευγνώμων προς την Επιτροπή που με επέτρεψε να συντάξω την έκθεση και να ξεκινήσω αυτό τον ε, διάλογο. Ευχαριστώ. Ο κύριος Αρσένης έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Όντως ο ανθρακάς είναι κάτι που δεν έχουμε εξετάσει και είναι πολύ σημαντικό Είναι ε, ατυχές που δεν έχουμε κάνει μία έκθεση για τον άνθρακα, αλλά εδώ μιλάμε για τα φράγματα, οπότε περιλαμβάνουμε και πολλά άλλα θέματα. Βρήκα όμως ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον ε, πώς ε, εντάχθηκε ο άνθρακας και τα καυσόξυλα στα φράγματα και καταλήξαμε στις πλημμύρες. Πάλι για ε, πλημμύρες. πρέπει να τονίσουμε τις παγκόσμιες προσπάθειες ε, ενάντια των κλιματολογικών αλλαγών θα πρέπει αυτό να τονιστεί περισσότερο και συμφωνώ για το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης. Υπάρχουν πολλές χώρες. Η Ιαπωνία είχε εξαιρετική, εξαιρετικό μηχανισμό έγκαιρης προειδοποίησης για το παλιριακό κύμα, αλλά ε, δεν προέβλεπαν τόσο τεράστιο. Και συμφωνώ ότι θα έπρεπε να καταρτήσουμε κάτι διαφορετικό. Να έχουμε δηλαδή ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης παγκόσμιο για τις χώρες που δεν μπορούν να το χρηματοδοτήσουν και δεν μπορούν να αποφύγουν τέτοιες καταστροφές. Έχω πολλές ιδέες σχετικά με το θέμα αυτό, αλλά θα σταματήσω εδώ προς το παρόν και στηρίζω στην ε, ανάγκη για κινήσεις για τον άνθρακα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ τον κύριο Ντέβα ο οποίος ανέλαβε να ε, ασχοληθεί με αυτό το πολύ σημαντικό θέμα και εγώ θα ήθελα πολύ να στηρίξω την ε, ε, ε, την εξέταση του άνθρακα και των ε, καυσόξυλων διότι είναι ένα θέμα που δεν έχουμε εξετάσει επαρκώς μέχρι στιγμής και το, Ευρωπαϊκό, το Παγκόσμιο Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για την Ανάπτυξη έχει καταρτήσει μια ομάδα εμπειρογνωμόνων για να για να εξετάσουν αυτό το θέμα και δημοσίευσαν πρόσφατα μία έκθεση η οποία διατυπώνει πολλές προτάσεις για να μειώσουμε αυτές τις επιπτώσεις και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ένα ρόλο να παίξει ε, για όλα τα θέματα που παρουσιάζονται στην έκθεση αυτή ε, και στον διάλογο με τις υποανάπτυξη χώρες. Θα μπορούσα ε, να μιλήσω για καθαρούς φούρνους για ψήσιμο, για καλύτερη χρήση φίλτρων, ε, για τα απόβλητα, ε, για την διαχείριση των αποβλήτων και άλλα. Είναι όλα θέματα που πρέπει να εξετάσουμε. Ο τίτλος αυτής της εκθέσεως είναι ίσως κάποιος μπερδεμένος. Υπάρχει το θέμα των φυσικών φραγμάτων που πρέπει να ε, ε, στηριχθεί και έχουμε και τα φράγματα τα οποία δημιουργούμε για άρδευση, για παραγωγή, για δικούς μας σκοπούς. Μην ξεχνάμε λοιπόν ότι το θέμα αυτό μπορεί να παρανοηθεί. Και θα ήθελα να τονίσω ότι η Ανεξάρτητη Επιτροπή ε, επίσης έχει δραστηριοποιηθεί και ίσως θα μπορούσε να όλοι, ε, ε, όλες αυτές οι επιτροπές να αναφερθούν στην έκθεση για να διατυπώσουμε κατευθυντήριες γραμμές για την κατασκευή των φραγμάτων διότι νομίζω ότι εμείς σαν πράσινοι θα θέλαμε να διατυπώσουμε μία τροπολογία ότι η Παγκόσμιος Τράπεζα θα πρέπει να σέβεται τα κριτήρια και τις ε, υποδείξεις της Παγκοσμίου ε, Επιτροπής για τα φράγματα. Ευχαριστώ. Τον λόγο έχει τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που εκπροσωπείται από τον κύριο Κόλλετ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον κύριο Ντέβα που συνέταξε αυτή την ε, έκθεση. Η έκθεση περιγράφει την αυξανόμενη απειλή που είναι νέα στο γενικό πλαίσιο των συζητήσεων σε διεθνές επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προφανώς έχει επίγνωση της νέας απειλής κυρίως στην περιοχή των Ιμαλαίων που αναφέρατε, αλλά και στη Λατινική Αμερική, στις Άνδης. Σε αρκετές χώρες, σε αρκετές περιοχές κινδυνεύουν από αυτό το ενδεχόμενο ε, τις πλημμύρες που προκαλούνται από την ταχεία τήξη των παγετώνων. Τώρα, όσον αφορά την πρόταση που κάνατε, που προτείνατε κάτι να γίνει στο πλαίσιο του ΟΗΕ, πιστεύουμε ότι υπάρχει δυνατότητα στο εφιστάμενο πλαίσιο. Η σύμβαση την αλλαγή του κλίματο αναφέρθηκε. Υπάρχει και ένα πλαίσιο για την αντιμετώπιση των καταστροφών, μείωση των κινδύνων για καταστροφέ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν δραστηριοποιηθεί σε αυτούς τους τομεί. και είμαστε έτοιμοι να προωθήσουμε το θέμα αυτό των νέων απειλών στην ε, διεξαγόμενη συζήτηση όσον αφορά τη μείωση κινδύνου καταστροφών. Υιοθέτησε Ευρωπαϊκή Επιτροπή Στρατηγική για την υποστήριξη μείωση των κινδύνων αυτών στις αναπτυσσόμενες χώρες και προσπαθούμε εκεί να καλύψουμε αυτά τα θέματα σαν βασικό στοιχείο αναπτυξιακής στρατηγικής τη μείωση των κινδύνων από φυσικές καταστροφές. Θέλουμε διάλογο, περιφερειακή προσέγγιση που προτείνατε και για τα Ιμαλάια, ένταξη των ανησυχιών σε εθνικές αναπτυξιακές στρατηγικές και στις περιφερειακές αλλά και συντονισμό μεταξύ των διαφόρων πρωτοβουλειών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως που ε, καλύπτουν αυτά τα ζητήματα. Ακριβώς λοιπόν για την Ασία και τη Λατινική Αμερική δεν έχουμε για την ώρα ειδική πρωτοβουλία για τη μείωση του κινδύνου φυσικών καταστροφών και πρέπει να συμπεριληφθεί στα έγγραφα για τη στατική για κάθε χώρα είναι ενταχθεί αυτή η πτυχή σε σφαιρικά προγράμματα, παγκόσμια προγράμματα. Ένα άλλο τομέας που μπορεί να καλύψει το ζήτημα που αναφέρατε είναι η συνεργασία για βιώσιμη διαχείριση των υδάτων. Αναφέρθηκαν τα φράγματα. Πιστεύουμε ότι πράγματι πρόκειται περί κρισίμου ζητήματος προς επίλυση αλλά όχι σαν ειδικό, ξεχωριστό. Καλύτερα να αντιμετωπιστεί στη σφαιρική προσέγγιση για τη διαχείριση των ε, χώρων ε, με τα ποτάμια και τα σημεία ε, συρροής υδάτων και ίσως τα πλαίσια θα πρέπει να επικαιροποιηθούν και η περιφερειακή συνεργασία είναι βασικό στοιχείο του όλου πλαισίου και θα πρέπει να υπάρχει ετοιμότητα για τις πλημμύρες. Ήδη υπάρχουν σχετικά προγράμματα στα προγράμματα συνεργασίας. Τρίτος τομέας πολιτικών, η αλλαγή του κλίματος. Και εκεί μπορεί να καλυφθεί το θέμα που θίξατε. Προσαρμογή και θα συνδεθεί με τη διαχείριση των υδάτων των ποταμίων ε, και προσέγγιση κατά χώρα, ε, η προσέγγιση όσον αφορά τη διαχείριση των δασών, καύση βιοκαυσίμων και τα καύσιμα που χρησιμοποιούνται η καύση των ξύλων, των καυσοξύλων, δημιουργεί ε, την εκπομπή αυτών των μορίων άνθρακα, των σωματιδίων άνθρακα, να αλλάξει τα καύσιμα εκπομπέ από ντίζελ και από άλλα καύσιμα, θα πρέπει να συνεργαστούμε με διεθνεί εταίρου, ούτω ώστε να ξέρουμε ότι ε, και οι εταίροι μα θα ακολουθήσουν αυστηρότερη πολιτική όσον αφορά την αποφυγή εκπομπή αυτών των σωματιδίων και του τι καίνε. Να προσέχουν τι καίνε. Και ένα συγκεκριμένο μέσο είναι η Παγκόσμια Συμμαχία για την Αλλαγή του Κλίματος. Έχουμε ένα πρόγραμμα στο Νεπάλ στα πλαίσια αυτά, που εστιάζεται στην προσαρμογή. Και για το 2011 θα κινηθούμε και στο Μπουτάν. Οι επαφές μας με τις αρχές του Μπουτάν προς αυτή την κατεύθυνση κινούνται, ολοκληρωμένη προσέγγιση. Και πώς μπορεί να ε, αντιμετωπιστεί αυτή η απειλή της, ε, του σπασίματος των φραγμάτων που αναφέρατε. Μετά από πρώτες αντιπροσωπείας μας στην περιοχή, εξετάζει τον δεχόμενο συνεργασίας με το Ινστιτούτο που αναφέρατε εσείς στην παρουσίασή σας. Έχει ξεκινήσει, έχει δρομολογηθεί η εργασία, δύσκολο να αναφέρουμε κάποια αποτελέσματα, αλλά πιστεύουμε ότι ίσως πριν το καλοκαίρι να είμαστε σε θέση να έχουμε ένα τελικό στοιχείο, κάποια τελικά στοιχεία, κατάλογο θεσμεών, χωρών που θα μπορούσαμε να συμπεριλάβουμε στο πρόγραμμά μας του 2011 σχετικά με αυτό το θέμα. Και μέσω της συμμαχίας της παγκόσμιας συναλλαγή του κλίματος όλο και περισσότερο δημιουργούμε δεσμούς μεταξύ των στόχων, δηλαδή προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος και μείωση του κινδύνου για φυσικές καταστροφές. Αρχικά τα βλέπουμε αυτά σε ξεχωριστά ξεχωριστές παρεμβάσεις, ξεχωριστούς τομείς. Αλλά οι δεσμοί είναι ξεκάθαροι και θα πρέπει να υποστηρίξουμε τις χώρες αυτές να αναπτύξουν σφαιρικές στρατηγικές για να καλύψουν και τους κινδύνους από φυσικές καταστροφές και να ακολουθήσουν ευρύτερη προσέγγιση όσον αφορά την προσαρμογή που απαιτείται για να αντιμετωπιστεί η αλλαγή του κλίματος. Αυτά και ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ντέβα, για να κλείσουμε κυρία Πρόεδρε, ε, έχω εκπλαγεί ευχαρίστως από την υποστήριξη της οποίας έτυχα από τους λαλίσαντες. Όταν ξεκίνησα τη δουλειά, τότε με προσπαθήσαν να σταματήσουν Επιτροπή Περιβάλλοντος. Μου λένε είναι ακραία θέματα αυτά αναψησιακά. Πρέπει να προχωρήσουμε. Κάποιος στην Επιτροπή Περιβάλλοντος υποθέτει ότι θα ετοιμάσει κάποια γνωμοδότηση, δεν είναι. Ναι, ναι. Κάποιο από την Επιτροπή περιβάλλοντο μπορεί να έρθει μαζί μα σε αυτή την κοινή προσπάθεια. Γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτά τα θέματα να τα εξετάζουμε πριν συμβούν και να βρούμε λύσεις οι οποίες προβλέπουν, αποφεύγουν αντί να τρέχουμε μετά σαν αποκεφαλισμένα κοτόπουλα ψάχνοντας να βγάλουμε άκρη και να διθώσουμε προβλήματα που θα μπορούσαμε να είχαν προβλέψει και διορθώσει εκ των προτέρων. Ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που ηγήθηκε στον τομέα. Δεν είχα ιδέα εγώ ότι ήδη έχετε επιτεθεί, έχετε μπει στο θέμα, το σκεφτόσαστε, μιλάτε με τους ε, κατοίκους του Μπουτάν κλπ. Τις αρχές του Μπουτάν. Εγώ ενεθάρρυνα τους συναδέλφους στην Επιτροπή να υποβάλουν όσο δυνατόν περισσότερες τροπολογίες για την έκθεση. Θα τους ενθαρρύνω και θα κανονίσω, ούτως ώστε το προσωπικό μου, ο κύριος Ρόμπισον και ο κύριος Ράσελ να έρθουν να συνομιλήσουν με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να το κουβεντιάσουμε και να δούμε πώς μπορεί να γίνει πιο στέρεα και γερή η έκθεση και να ξεπεράσει την Ευρωπαϊκή Ένωση, να πάει και στα ΟΗΕ και αλλού και στις κυβερνήσεις αυτών των χωρών που φαίνεται να είναι σε άλλο πλανήτη να ζουν σχετικά με αυτά τα προβλήματα. Και να αρχίσουμε να τους κλωτσάμε λίγο, να τους ταρακουνάμε για να κάνουν κάτι. Χαίρομαι λοιπόν που έτυχα αυτής της ε, υποστήριξης. Ευχαριστώ. Δεν σας είδα, έχετε το λόγο. Ε, ευχαριστώ. Θα ήθελα να θέσω το θέμα των, των προθεσμιών για τις τροπολογίες. Λέει στο πρόγραμμα 24 Μαρτίου, αλλά ανεβλήθη έτσι. Εκτός, εκτός μικροφώνου. Άλλαξαν τα πράγματα, λέει πρόεδρος. Η ημερομηνία που θα σας έλεγα είναι 11 Απριλίου, 12 το μεσημέρι. Μέχρι τις 11 Απριλίου έχουμε χρόνο, το μεσημέρι λοιπόν, και η έκθεση θα ψηφιστεί στις, στις 25 Μαΐου. Θα ξεκινήσουμε τώρα, θα περάσουμε στο σημείο 18 της ημερήσιας διάταξης. Λοιπόν, η ΚΑΠ στον ορίζοντα 2011 διατροφή, φυσική πόρη, η ύπεθρος και πώς θα αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις του μέλλοντος. Είναι θέμα πολύ σημαντικό για το μέλλον της κοινή αγροτικής πολιτικής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε μέσα Νοεμβρίου μια ανακοίνωση που αποτέλεσε αντικείμενο εκθέσεως πρωτοβουλίας που προετοίμασε η Επιτροπή Γεωργίας. Ο συνάδελφός μας Κρήτον Αρσένης είναι εισηγητής της Επιτροπής Ανάπτυξης η σύνταξη της γνωμοδοτήσεώς μας επί της εκθέσεως της Επιτροπής Γεωργίας. Ο κύριος Αρσένης, έχετε το λόγο λοιπόν για να παρουσιάσετε την γνωμοδότησή σας. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Πολύ λίγοι είμαστε στην αίθουσα. Θα προσπαθήσω λοιπόν να είμαι πολύ σύντομος. Γνωρίζουμε πόση σωρευτική αρνητική συνέπεια έχει η ΚΑΠ σε αναπτυσσόμενες χώρες. Στην ΚΑΠ υπήρξαν κάποια θέματα τα οποία δεν είναι επιζήμια, αλλά σιγά σιγά μέσω των διαφόρων μεταρρυθμίσεων άλλαξαν τα πράγματα και υπάρχουν ε, επιβλαβείς επιπτώσεις, αρνητικές. Θα πρέπει λοιπόν να γίνει στην ΚΑΠ πρόνοια ώστε να μην υπάρχουν τέτοιου είδου αρνητικές συνέπειες για τις αναπτυσσόμενες χώρες. Κατά τον σχεδιασμό της λοιπόν θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί ώστε να μην δημιουργούμε προβλήματα στον κόσμο, ανά τον κόσμο. Αρχίσαμε ε, ζητώντας να καταργηθούν οι επιδοτήσεις εξαγωγές κάποιες από τις επιδοτήσεις προβλέποντας τα πλαίσια των ανταλλαγών με διάφορες συμφωνίες που είχαμε με χώρες, φαίνεται ότι θα πρέπει να προβλέψουμε μεταβατικές καλλιέργειες για να μπορέσει σιγά σιγά να σταματήσει τις εξαγωγικές επιδοτήσεις η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι άλλο πρέπει να κάνουμε. Τα τραύματα που δημιουργήσαμε να μπορέσουμε να τα θεραπεύσουμε. Η ΚΑΠ δεν είναι μια πολιτική που μπορεί να έχει μέτρα που επηρεάζουν άμεσα άλλες χώρες. Τι μπορεί να κάνει όμως. Αντί να δημιουργήσουμε, για να βελτιώσουμε την κατάσταση, να χρησιμοποιήσουμε την αναπτυξιακή μας πολιτική και άλλες πολιτικές για την ε, ασφάλεια των ειδών διατροφής ε, κάποιων ε, χωρών, να εξαλείψουμε τα φαινόμενα διαρπαγής γης, να εξασφαλίσουμε τα ιδιοκτησιακό καθεστώς μικροκαλλιεργητών και ηθαγενών καλλιεργητών, να εξασφαλίσουμε πρόσβαση σε σπόρους και να μην ε, υποβάλλουμε τους πάντως εξάρτηση από παρασιτοκτόνα. Κάτι άλλο το οποίο θα πρέπει επίσης να προσέξουμε είναι η κερδοσκοπία. Δεδομένου ότι δεν υπάρχει μόνο κερδοσκοπία στον ε, οικονομικό τομέα, αλλά και στα είδη διατροφής. Διότι υπάρχουν ε, βασικά αγαθά των οποίων η τιμή αποτελεί σημείο εκμετάλλευση. Θα αναφέρω τα σιτηρά, Θερυπίν. Θα πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε πώς θα αντιμετωπίσουμε και την ε, κερδοσκοπία που παρατηρείται και ε, εντό της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης, να δούμε πώς θα μπορέσουμε να κάνουμε τις συναλλαγές μας στις διάφορες αγορές. Και επίσης, τι θα κάνουμε με την ε, Διεθνή Εμπορική Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Μερκοσούρ, της χώρας Μερκοσούρ λοιπόν της Λατινικής Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όποιος έχει δει την μελέτη αξιολόγηση των επιπτώσεων της Επιτροπής, θα έχει παρατηρήσει ότι πρόκειται για μια πολύ κακιά συμφωνία και για το περιβάλλον και για την γεωργία αυτών των χωρών. Ε, πρόκειται για μια πολιτική που καταστρέφει μεγάλες περιοχές του Αμαζονίου εκεί αναπτύσσονται και διάφορες παράνομες ενέργειες ε, ε, υλοτομίες, παράνομες ενέργειες στην καλλιεργήσιμη γη και κίνδυνοι και για τους καλλιεργητές αλλά και για την κοινωτική γεωργία. Αυτές ήταν οι κυρίες παρατηρήσεις μου και αναμένω με ενδιαφέρον τις παρατηρήσεις των συναδέλφων. Η κυρία Κέλλερ, ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την έκθεση αυτή που την χαιρετίζουμε ως πράσινη. Έχουμε ε, κάποια περιορισμένη όρια, αλλά μπορούμε με την κατάθεση τροπολογιών να προσθέσουμε κάποια στοιχεία. Θα θέλαμε να αναφέρεται περισσότερο η αναπτυξιακή πολιτική. Η... Κάποιες θα πρέπει να υπάρχουν νομοθετική πράξη πέρι μεταρρύθμιση της ΚΑΠ. Είπαμε ότι δεν θα πρέπει μόνο όπως λέγει η παρούσα πρόταση να διαφορόμαστε μόνο από τις τους τρόπους παραγωγής. Θα θέλαμε επίσης να γίνει αναφορά στις ε, κλιματικές αλλαγές και την επιρροή της ε, γεωργίας που ευθύνεται για τις εκπομπές ε, για, το φαινόμενο θερμοκηπίου σε ποσοστό 40%. Το όλο θέμα στη ζήτηση που γίνεται είναι να μην περιοριστούμε σε αυτά τα οποία λέμε εδώ στην Επιτροπή Ανάπτυξης, διότι καλά τα λέμε όλα αυτά, αλλά θα πρέπει οι ιδέες μας να μπορέσουν να περάσουν και στην Επιτροπή Γεωργίας, που είναι η Επιτροπή η οποία γινόταν των συζητήσεων που γίνονται και το υπεύθυνη για τα, και επί υπεύθυνη για όλες τις νομοθετικές πράξεις που οδηγήσουν και στις αλλαγέ της ΚΑΠ. Το... οι γνωρίζει, δεν μπορεί να μην γνωρίζουμε ότι η δική μας κοινή αγροτική πολιτική δεν έχει επιπτώσεις ανά τον κόσμο. Θα πρέπει λοιπόν μεταξύ της Επιτροπής Γεωργίας και της δικής μας να υπάρξει ε, κάποια ε, διασύνδεση. Να μην κάνουμε χωριστά κάποια πράγματα. Θα πρέπει να καλέσουμε κάποιους ε, συναδέλφους της ΚΑΠ να μιλήσουμε για θέματα σημαντικά, όπως αυτό που θα κάνει την ακρόαση του Ιουνίου, τα θέματα της ασφάλειας των ε, ειδών διατροφής. Και παραλαμβάνω ότι κάνουμε δεν θα πρέπει να περιορίζεται στους τείχους αυτής της αίθουσας στην οποία συνεδριάζουμε. Θα πρέπει ό,τι κάνουμε και ε, ό,τι κάνει η Επιτροπή Ανάπτυξης να ακουστεί και να εισακουστεί από την Επιτροπή Γεωργίας. Ευχαριστώ. Τώρα για την ε, Επιτροπή η κυρία Μοτερό. Όχι. Α, ευχαριστώ. Ε, εγώ θα μιλήσω εν ονόματι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, θα... θα αναφερθώ σε τέσσερα σημεία μεταξύ των πολλών της γνωμοδότησης αυτής της Επιτροπής. Καταρχήν ε, της επίπτωσης της κοινή γεωργικής πολιτικής στις υποανάπτυξη χώρες, το θέμα της ε, διατροφικής ασφαλείας σε σχέση με την γεωργία, την κερδοσκοπία και την ρύθμιση του ε, αγοράς ε, των παραγόγων προϊόντων και τοπικών προϊόντων και τις ανταλλαγές ε, με τις χώρες του Μερκοσούρ. Το άρθρο 208 της Συνθήκης συζητά από την Ευρωπαϊκή Ένωση να λάβει υπόψη την αναπτυξιακή ε, συνεργασία, ιδίω όσο αυτό, αυτή επηρεάζει τις υποανάπτυξη χώρες και ε, στο θέμα αυτό υπάρχει η αρχή της αποφυγής βλαβών που ανέφερε ο κύριος Αρσένης. Στα, πλαίσια αυτά και σύμφωνα με τις δεσμεύσεις για καλύτερη ρύθμιση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτή τη στιγμή προβαίνει σε μία ανάλυση επιπτώσεων για να μπορέσει να εξετάσει τις αποφάσεις που άπτονται της γεωργικής πολιτικής και εξετάζει και τις ε, εμπορικές σχέσεις με τις υποανάπτυξης χώρες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ευχαρίστως ε, θα ενημερωνόταν για τα στοιχεία στα οποία βασίζεται η αξιολόγηση των αρνητικών επιπτώσεων της ε, κοινή της γεωργικής πολιτικής ή στις υποανάπτυξη χώρες, διότι εμείς ε, όλο και περισσότερο δυσκολευόμαστε να μπορέσουμε να επαληθεύσουμε αξιόπιστα τις, τις για αρνητικές επιπτώσεις υπό ανάπτυξη χώρες, διότι ε, μία διαδικασία αναθεωρήσεω που έχει ξεκινήσει το 1992 λέγει ότι η στήριξη της ε, ευρωπαϊκής ε, γεωργίας στην εποχή όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση επηρέαζε την πολιτική τιμών ε, έχει περάσει. Τώρα έχει αλλάξει η κατάσταση και οι, ε, οι ενδιαφερόμενοι υφίστανται τις τιμές που, διοργανώνουν, που διαμορφώνουν οι αγορές. Οπότε πρέπει να γίνει μία ανάλυση επιπτώσεων μέχρι το 2020 για να εξετάσουμε και την ε, το αποτελέσμα της μειώσεως της ευρωπαϊκής ε, πολιτικής ε, πολιτικής παραγωγής και της αυξήσεως των εισαγωγών. Όσον αφορά τη στήριξη των ε, εισαγωγών, νομίζω ότι είναι πρόθεση Ευρωπαϊκής Ένωσης να τις μειώσει από το 2003 βάσει αμοιβαιότητος ε, με τις χώρες του ΟΣΑ. Ε, συνδεδεμένες με αυτή την ε, αντιμετώπιση και για να αντιμετωπίσουμε την αυξανόμενη ζήτηση η κοινή οργική πολιτική θέλει να διατηρήσει τη δυνατότητα παραγωγής ακόμη και όπου δεν προσφέρονται συνθήκες και η γεωργία είναι αναγκαία για να υπάρξουν περιβαλλοντολογικά δημόσια αγαθά ή όπου καθορίζει τις ισορροπίες μεταξύ των περιφερειών. Έτσι θα συμβάλλει ε, σε δύο ουσιαστικά θέματα, καταρχήν αποφεύγοντας τη στρέβλωση ε, των ε, των συνθήκων αναπτύξεων των υποανάπτυξης χωρών και Υπάρχουν συγκεκριμένες ενέργειες στην διατροφική αλυσίδα η οποία θα επηρεάσει ε, τις, ε, ε, ε, τις εξελίξεις και αυτά όλα αυτά θα ξαναεξεταστούν στο τέλος του χρόνου. Θέλουμε επίσης να εξασφαλίσουμε και την, την τροφοδότηση της αγοράς και όσον αφορά τις τοπικές αγορές θα πρέπει οι εντόπιοι παράγοντες να γνωρίζουν πώς μπορούν να εξυπηρετήσουν καλύτερα τα συμφέροντά τους. Αλλά βασιζόμαστε εις ε, την ε, τοπική τροφοδότηση για την ε, διατροφική αλυσίδα και σήμερα πρέπει οι γεωργοί να αντιμετωπίζουν και τους κινδύνουν βάσει με και μέτρων τα οποία αναθεωρούμε αυτή τη στιγμή στα πλαίσια της γενικότερης αναθεώρησης. Οι σχέσεις με το Μερκουσούρ έχουν αξιολογηθεί επανειλημμένως. Έγινε ένα sustainability impact assessment από εξωτερικούς συνεργάτες που είναι και είναι οι πιο πλήρεις από αυτές τις αξιολογήσεις με στόχο να αξιολογήσουμε τις δυνατότητες και τις επιπτώσεις της συμφωνίας για να μπορέσουμε να αναλάβουμε τις δέουσες πρωτοβουλίες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τοποθετήθηκε βάσει αυτής της αξιολόγησης, δημοσίευσε την θέση της μαζί με την αξιολόγηση. Αυτή, αυτό το έγγραφο ε, αναμορφώνεται και ενημερώνεται και θα περιλάβει και τη γεωργία στην ε, ανάλυση επιπτώσεων των ε, μεταρρυθμίσεων. Αυτές ήταν ορισμένες παρατηρήσεις τις οποίες ήθελα να κάνω σχετικά με ορισμένα σημεία της γνωμοδότησης που συζητάτε. Ευχαριστώ. Κύριε Αρσένη, έχετε το λόγο τώρα για να καταλήξετε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όσον αφορά τις εξαγωγικές επιδοτήσεις, με τα σας άκουσα ότι... Μάλλον είδα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν τις έχει εξαλείψει, δεν είναι ξεκάθαρο. Δεν είναι τίθετο θέμα να παραμείνουν εξαγωγικές επιδοτήσεις. Έλεγε ότι όλοι πρέπει να κινούνται σε ισότιμη βάση, έλεγε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν υπάρχει σαφής σχέσεις μεταξύ αυτών που είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξαγωγικέ ε, Επιδοτήσεις και τις, με την ασφάλεια τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, στην έκθεσή μου αναφέρω ότι έχει μειωθεί ο αντίκτυπος, σημαντικά οι αρνητικές συνέπειες, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν συνέπειες και δεν είναι ξεκάθαρο τι έχουμε κάνει. Ας μας πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι κάναμε για να γιατρέψουμε τα τραύματα, τις πληγές που ανοίξαμε. Είπαμε τώρα ότι ο αντίκτυπος είναι πολύ μικρότερος. Τι κάναμε για να αποκαταστήσουμε τις βλάβες που προξενήσαμε. Αυτό προσπαθεί να καλύψει η έκθεση. Κυρίω μέσω τη συνοχή τη πολιτική που ακολουθούμε και τη εμπορευματική και αναπτυξιακή μα πολιτική, εάν δεν μπορεί να αναλάβει δράση η κοινή αγροτική πολιτική εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση. Για τι συμφωνίε Μερκοσούρ, Ευρωπαϊκή Ένωση Μερκοσούρ, με συγκλώνησαν τα σχολεία σα, θα έλεγα. Όταν μιλάμε για την αποδάσωση 11% των δασών των τροπικών του Αμαζονίου, δεν είναι ακόμα μια συνέπεια αυτή με την οποία θα πρέπει να ασχοληθούμε. Αν αυτή είναι η προσέγγιση σας, ουε. Έχουμε τεράστια απόσταση μεταξύ μας στις προσεγγίσεις. Θα ήθελα να πω ότι δεν είναι στοιχείο που μου έδωσε μη κυβερνητική οργάνωση. Ήταν από την αξιολόγηση βιωσιμότητας ε, που αναφέρεται στο, στο ποσοστό της αποψήλωσης των δασών. Είναι χρήματα που έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ανεξάρτητο φορέα για να κάνει αυτή την αξιολόγηση. Από εκεί προέρχεται αυτό το στοιχείο και δεν είναι μικρό νούμερο. 11% του Αμαζονίου, των δασών του Αμαζονίου. Γι' αυτό μιλάμε. Η αξιολόγηση έγινε όχι για να δούμε τι συνέπειες της συμφωνίας, αλλά για να δούμε τι πρέπει να αλλάξουμε στη συμφωνία. Να μην αρχίσουμε να προετοιμαζόμαστε για τις ε, συνέπειες, να αποφύγουμε τη ζημιά. Και ελπίζω αυτό το μήνυμα να είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο για την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Λοιπόν, λέει η Πρόεδρος, έχουμε μέχρι τις 28 Μαρτίου, μεσημέρι 12, προθεσμία υποβολή τροπολογιών, ψηφοφορία, στις 13 Απριλίου. Νομίζω ότι είναι μια συζήτηση που διαρκεί σειρά ετών, είναι αργά, έχετε δίκιο, ουσιαστικά για να φύγουμε από ένα διάλογο που καμιά φορά είναι διάλογος κοφών, θα πρέπει να δούμε συγκεκριμένα ποιες συνέπειες. Στις αναπτυσσόμενες χώρες να αμφιζητήσουμε τις επιδοτήσεις δεν είναι αυτό το θέμα. Είναι οι αλλαγέ οι οδυνηρέ. Η δημόσια πολιτική που αλλάζει. Τι συνέπειε έχει. Όσον αφορά τη φτώχεια, την ασφάλεια, τη διατροφική κλπ. Οι αλλαγέ οφείλονται στην αγροτική πολιτική, στην εθνική πολιτική. Από εκεί εξαρτώνται από την αναπτυξιακή πολιτική, την εθνική. Εξαρτάται τις επενδυτικέ πολιτικές των μεγάλων ε, εταιριών τροφίμων από την πτυτικότητα των δημών των πρώτων υλών. Αν το πιάσουμε αυτό δεν τελειώνουμε. Τι προσπαθούμε να κάνουμε. Να έχουμε μια αξιολόγηση συγκεκριμένη, στέρεη, όσον αφορά την επιστημιστική ασφάλεια. Δεν διατηνόμαθα ότι το θέμα αυτό σε παγκόσμιο επίπεδο αφορά την κοινή αγροτική πολιτική. Υπάρχει πρόσφατη ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που προτείνει στατηγικό πλαίσιο της Ένωσης για να βοηθηθούν αναπτυξόμενες χώρες να αντιμετωπίσουν την πρόκληση αυτή που έχουν όσον αφορά την επιστημιστική ασφάλεια. Προσπαθούμε να ταιριάξουμε διάφορα εργαλεία που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να αντιμετωπιστεί αυτή η πρόκληση. Τα περισσότερα εργαλεία είναι εκτός της κοινή αγροτικής πολιτικής για την αποδάσωση, για τον ψήφιση των δασών, κανείς δεν το αρνιέται. Υπάρχει πραγματικός κίνδυνος. Είναι πραγματικός ο κίνδυνος. Και είναι οι χώρες, οι χώρες του Μερκοσούρ είναι χώρες που δεν έχουν υπογράψει τη συμφωνία του Κιώτο. Δεν υπέχουν καμία υποχρέωση μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου. Είναι προφανές. Αν υπάρχει μετακίνηση της παραγωγής υπάρχει πραγματικός κίνδυνος για τις αλλαγές του κλίματος. Κανεί δεν το αρνείται. Δεν το αρνούμεθα σαν πτυχή. Τοποθετήθηκα επί της ΚΑΠ και του ρόλου που έχει. Μάλλον να το κάνω αυτό, ε, δεν βλέπω πώς μπορεί να συσχετιστεί η ΚΑΠ με αυτό το φαινόμενο, αυτό το κίνδυνο. Για να επανέλθω στο πρώτο σημείο που ανέφερε ο εισηγητής. Συγκεκριμένες περιπτώσεις. όπου οι αλλαγές της ΚΑΠ έχουν ως αποτέλεσμα να επηρεαστούν, να πληγούν ευάλωτοι πληθυσμοί σε αναπτυσσόμενες χώρες. Είναι ένα πραγματικό ειλικρινές ερώτημα αυτό. Δημιούργησε διεύθυνση. Τη διεύθυνσή μου Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πάντα στρέφεται προς την αρμόδια διεύθυνση και τις διευθύνσεις που έχουν εκπροσώπους αναπτυσσόμενες χώρες για να ζητήσουν να δουν αυτό, να διαπιστώσουν αυτό, κατά πόσο εξαγωγικές επιδοτήσεις πληρούν τις προϋποθέσεις και οι χώρες συμμορφώνται με τις υποχρεώσεις. Οι εξαγωγικές επιδοτήσεις μετά από 15 χρόνια μειώθηκαν. Δεν έχω στοιχεία συγκεκριμένα μειώθηκαν δραματικά. Δεν υπάρχουν σχεδόν. Ξαναχρησιμοποιήθηκαν εδώ και δύο χρόνια, τη στιγμή της κρίσεως των γαλακτοκομικών προϊόντων. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μελέτη για να δούμε κατά πόσο είχε αντίκτυπο σε κάποια αναπτυσσόμενη χώρα αυτό. αυτή η προσωρινή αποκατάσταση των εξαγωγικών ε, επιδοτήσεων σε μια περίοδο κρίσης. Κατά πόσο είχαν συνέπειες, είχε συνέπειες σε αναπτυσσόμενες χώρες. Ευχαριστώ. Θα σε έδωσα την τροπολογία. 28 Μαρτίου, μεσημέρι, 12 το μεσημέρι, για τις τροπολογίες, λέει Πρόεδρος. Έχουμε ακόμη ένα θέμα στην ημερήσια διάταξη που είναι η ενημέρωση για την ε, παρακολούθηση των εκλογών στην Ουγγάντα. Είναι πολύ βασικό θέμα και νομίζω ότι είναι κρίμα σε αυτή η παρουσίαση να γίνει τόσο αργά με τόσο λίγους παρόντες. Αποφάσισα λοιπόν να ε, αναβάλω το θέμα αυτό για μια επόμενη συνεδρίαση, ε, στην επόμενη συνεδρίασή μας και ε, θα ήταν καλύτερο να μπορέσουν όλοι να ακούσουν τι γίνεται. Η επόμενη συνεδρίασή μας λοιπόν θα γίνει 12 Απριλίου στις Βρυξέλλες από τις 15 έως 18 και 30 και 13 Απριλίου 9 ε, 12.30 και 3 ε, με 6.30 το απόγευμα. Λύεται η συνεδρίαση